Good morning everybody. Καλημέρα σας. Κυρία Πρόεδρε Καριεντζέβα, κύριε Αντιπρόεδρε Ντομπρόφσκης, ε, μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, συνάδελφοι του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι μεγάλη μου χαρά να σας βλέπω εδώ συγκεντρωμένους για αυτή την πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας. είναι η μεγαλύτερη διακοινοβουλευτική εκδήλωση στο πρόγραμμά μας. Η πρωτοβουλία αυτή. Φέτος 123 μέλη από 27 ευρωπαϊκές χώρες και 56 κοινοβουλευτικές 56 ε, βουλές έχουν συγκεντρωθεί εδώ. Εκπροσωπούνται και η Νορβηγία και η Ελβετία μεταξύ μόν. Τα εθνικά κοινοβούλια παίζουν καθοριστικό ρόλο ώστε οι ευρωπαϊκές πολιτικές να είναι πιο κοντά στους πολίτες. Και αυτό είναι καθοριστικό και για τη δική μου τη θητεία ω Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να βρούμε τρόπου να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ένωσή μα και τα θεσμικά τη όργανα. Πρέπει να προσφέρουμε ένα νέο όραμα για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να προτείνουμε συγκεκριμένη δράση που να είναι δίκαιη και σωστή για την Ευρωπαϊκή Ένωση προ όφελο όλων τα ερχόμενα χρόνια. Για να το πετύχουμε αυτό, το Ευρωκοινοβούλιο θεωρεί ότι η διακοινοβουλευτική συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κοινοβουλευτικών συνελεύσεων είναι ζωτική σημασίας για να χτίσουμε μαζί το μέλλον της Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μου να συνεχίσω στη μητρική μου γλώσσα. Τις δύο αυτές ημέρες συζητούμε την αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών στην Ευρώπη των πολιτικών ανάπτυξη, σταθερότητα και οικονομική διακυβέρνηση. Η οικονομική ανάπτυξη, ανάκαμψη στην Ευρώπη μετά από 10 χρόνια κρίσης είναι βεβαίως καλή είδηση. Ωστόσο βλέπουμε ότι η ψαλίδα μεταξύ φτωχών και πλουσίων, ε, προηγμένων και καθυστερημένων περιοχών μεγαλώνει. Το 80% του νέου πλούτου πηγαίνει μόνο στα χέρια του 15% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Αυτή η ασυμμετρική ανάπτυξη δεν προσφέρει αρκετές ευκαιρίες εργασίας, ιδίως για τους νέους. 23 εκατομμύρια άνθρωποι μεταξύ των 15 και 23 δεν φοιτούν πουθενά και δεν εργάζονται. Η μέση τάξη πάντοτε φοβάται, ακόμα περισσότερο μάλλον φοβάται από ποτέ την οικονομική υπαναχώρηση. Οι νέες γενιές έχουν χειρότερες ε, προσδοκίες και προοπτικές από ότι οι γονεί τους. Τα χρόνια αυτά η παγκόσμια οικονομία έχει ακολουθήσει παρόμοιε τάσει. Η τεχνολογική ανάπτυξη, η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και ακόμα ανοιχτότερε αγορέ βεβαίω επέτρεψαν την οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, αλλά δημιουργήσαν και ανταγωνισμό ε, προ ε, τα για τον, ε, με το φορολογικό ανταγωνισμό οι μεταναστευτικέ ροέ που πολλέ φορέ είναι ανεξέλεγκτε και το φθηνό εργατικό δυναμικό έχουν πλήξει κυρίω τι πιο αδύναμε ομάδε του πληθυσμού που έχουν να αντιμετωπίσουν την απογοήτευση του αποκλεισμού και τη της κοινωνική δυσφορία. Το μόνο αποτελεσματικό όπλο κατά τη δυσαρέσκεια αυτή είναι χειροπιαστέ αποκρίσει που μόνο μια ενωμένη Ευρώπη, πιο δημοκρατική Ευρώπη και πιο αποτελεσματική μπορεί να προσφέρει. Μόνο εάν εργαστούμε όλοι μαζί μπορούμε πραγματικά να, φέρουμε, να κάνουμε διαφορά σε θέματα που έχουν ε, σημασία διακρατική, αφορούν όλα τα κράτη και τον δικό μας ρόλο ως φορέα μπορούν να επιτρέψουν να τον ασκήσουμε απέναντι γιγάντων ε, της οικονομίας όπως ε, η ΕΠΑ, ΕΕ, η Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία. Η πρόκληση που έχουμε μπροστά μα είναι διπλή. Δεν αρκεί να ενισχύσουμε την ανάπτυξη τη οικονομία, αλλά πρέπει να φροντίσουμε η ανάπτυξη αυτή να φέρει κέρδη και για ε, και ελπίδε κερδοφορία για μεγαλύτερο μέρο του πληθυσμού. Μόνο έτσι θα είμαστε συνεπεί με τι θεμελιώδει αξίε μα. Ελευθερία και ανθρώπινη εξωπρέπεια. Και μέσω τη εργασία η τεχνολογική επανάσταση, η ψηφιακή επανάσταση, η ρομποτική, η τεχνητή ευθεία μεταμορφώνουν πλήρως τον κόσμο της εργασίας και της απασχόλησης. Πρέπει οι ευρωπαϊκές πολιτικές να παρακολουθήσουν αυτές τις εξελίξεις, υποστηρίζοντας όχι μόνο τις προσπάθειες των εταιριών και επιχειρήσεων, αλλά και των εργαζομένων με τεράστιες επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, που να ευνοούν την προσαρμογή των δεξιοτήτων τους στις νέες απαιτήσεις. Πρέπει επίσης να χειριστούμε και την τεχνολογία με ψηφιακές πλατφόρμες. Ένας γίγαντας του διαδικτύου, ε, μια μεγάλη εταιρεία, δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη ως προς τους φόρους, την προστασία των προσωπικών ελευθεριών, την τήρηση δεδομένων και τους καταναλωτές. Πρέπει να υπάρχει ευημερία, να το προσφέρει αυτό η Ένωση με δικαιοσύνη και στα φορολογικά θέματα. Η ανάπτυξη και η ισότητα απαιτούν και την ολοκλήρωση του οικοδομήματος που ως τώρα έχουμε θέσει τα θεμελιά του με την εσωτερική αγορά και τον πυλώνα του ευρώ. Απομένουν όμως ακόμη πολλά να γίνουν. Η αγορά μας πρέπει να αναπτύξει όλες τις δυνατότητές της πολύ συχνά σε τομείς όπως οι υπηρεσίες, η ενέργεια, ε, τα ψηφιακά και ε, τα κεφάλαια, οι κεφαλαίοι αγορές. Αυτή η ένωση σημαίνει να ενισχύσουμε την εργασία, ...της μικρομεσαίας επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και να φροντίσουμε οι λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές να έρθουν πιο κοντά στην ανάπτυξη των πλουσιότερων. Η Ένωση των Κεφαλαιγορών και η Τραπεζική Ένωση μπορούν να προωθήσουν τη φορολογική σύγκληση, την οικονομική σύγκληση και την πολιτική. Δεν μπορούμε να έχουμε κοινό νόμισμα χωρίς να φτάσουμε σε πιο ε, ομοιόμορφα επίπεδα ανταγωνιστικότητας και οικονομική σύγκληση καθώς και κοινωνική σύγκληση συνολικότερα. Πρέπει να περιορίσουμε τους οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους, αλλά με κοινά εργαλεία για να μπορούμε να τους προλάβουμε. Το Κοινοβούλιο τον περασμένο Φεβρουάριο ενέκρινε τρεις εκθέσεις για να βελτιωθεί η οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης. Θέλουμε να υπάρξει ένα Υπουργό Οικονομικών Υποθέσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να, να διενεργήσει τι απαραίτητε παρεμβάσει για, την, για το χώρο τη εργασία και την οικονομία. Επίση, χρειάζονται περισσότερε δημόσιε επενδύσει, ε, κονδύλια και πόροι για την τεχνολογία και την ανάπτυξη, ώστε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί παγκοσμίω. Το Κοινοβούλιο επίσης ε, τέθηκε υπέρ της ε, μετατροπής του Ταμείου για τη διάσωση των κρατών σε ένα πραγματικό Ευρωπαϊκό Ταμείο ώστε να διορθώνονται οι κοινωνικές ανισότητες και να διευκολύνονται οι διορθωτικές μεταρρυθμίσεις. Τα εργαλεία αυτά απαιτούν μια οικονομική διακυβέρνηση που να είναι διαφανής και δημοκρατική. Γι' αυτό το Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και πρέπει να συνεργαζόμαστε πάντοτε εντατικά μεταξύ μας. Αυτήν την πρώτη χρονιά, από την πρώτη μάλλον χρονιά της Προεδρίας μου στο Κοινοβούλιο, έκανα ό,τι μπορούσα για να μπουν στο κέντρο όλων των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα θέματα αυτά ώστε να είμαστε ακριβώ ο χώρο που εκπροσωπεί του λαού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι το πρώτο θεσμικό όργανο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρόλο μα είναι να ελέγχουμε ε, τον, ε, την εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όχι μόνο να διαβάζουμε αυτό που μα έρχεται από τα μέγαρα που βρίσκονται εδώ γύρω μα, αλλά να εκπληρώνουμε πλήρω το ρόλο μα ω συνομοθετών. Και αυτό ε, σε πλήρη συμφωνία και συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει και αυτά να, να επεχρεπνούν και να παρακολουθούν το έργο μας, για να βλέπουν αν πάντοτε σεβόμαστε τους κανόνες της επικουρικότητας. Πρόκειται για μια συνεργασία πολύτιμη. Στο κέντρο της βρίσκεται ο πολίτης, το κέντρο κάθε πολιτικής δράσης, διότι αν το κοινοβούλιο, εάν τα κοινοβούλια χάσουν αυτό το ρόλο, χάνει το ρόλο του και ο πολίτης Χάνουμε την ουσία της δημοκρατίας. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι σε αυτή την δύσκολη στιγμή, την μετάβαση, όπου βλέπουμε να υπάρχουν τόσοι φόβοι στην Ευρώπη και νέες ευκαιρίες. Ε, η δουλειά λοιπόν που θα κάνει εδώ το Ευρωκοινοβούλιο, η δουλειά των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι ζωτική σημασία. Διότι τα κοινοβούλια είναι το σημείο σύνδεσης των πολιτών, των λαών με την εκτελεστική εξουσία. Δική μας δουλειά λοιπόν είναι πάντοτε να εργαζόμαστε προς όφελος των πολιτών. Ο στόχος της, εβδομάδας, της κοινοβουλευτικής αυτής εβδομάδας είναι ακριβώς αυτός. Να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή τα εθνικά κοινοβούλια. Τα δύο πάνελ που θα ακολουθήσουν είναι ένα παράδειγμα κοινή διακυβέρνηση. Το πρώτο θα επικεντρωθεί στο ρόλο που θα έπρεπε να έχουν τα κοινοβούλια στο μηχανισμό σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το επόμενο θα επικεντρωθεί στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την επόμενη περίοδο. Εδώ θα δούμε κατά πόσο ο προπολογισμό θα πρέπει να έχει πολιτική διάσταση για να αντιμετωπίσει τι πραγματικέ ανησυχίε των ε, πολιτών, την ε, ανεργία των νέων, την ε, λάθρομετανάστευση, τα εργαλεία για την άμυνα και την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Εάν ο κοινοτικό προπολογισμό παραμείνει απλώ ένα μηχανισμό ανακατανομή κονδυλίων, δεν θα πετύχει αν δεν έχει πολιτικούς στόχους. Πρέπει να προσφέρει προστιθέμενη αξία για να περάσουμε από την εποχή της κρίσης στο να δώσουμε καλύτερες αποκρίσεις στα προβλήματα των πολιτών. Η έγκριση των τριών εκθέσεων του Κοινοβουλίου, η υπογραφή της δήλωσης της Ρώμης 25 Μαρτίου του 2017 και οι δηλώσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξαν τη συζήτηση για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωκοινοβούλιο παρακολούθησε στενά όλη αυτή τη ε, δουλειά, ε, καλώντα όλου του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων να εκφραστούν στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Ακούσαμε τον ε, Πρωθυπουργό τη Κροατία και θα ακολουθήσουν ο Πρωθυπουργό τη Πορτογαλία και ο Γάλλος Πρόεδρο. Τον έχουμε διάλογο και να ανταλλαγή ιδεών στο σώμα μα είναι ακόμη ένα ενθαρρυντικό βήμα για να έχουμε μια ανοιχτή και διαφανή συζήτηση για τα θέματα αυτά. Και να επιτρέψουμε για άλλη μια φορά στο Ευρωκοινοβούλιο να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων για το μέλλον τη Ένωση. Δεν είναι μέλλον τη γραφειοκρατική διοίκηση. Είναι ε, συζήτηση για το μισό δι ανθρώπων, ανδρών και γυναικών που ζουν στα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε συζήτηση ανοιχτή ε, και ενίσχυση της δημοκρατικής διαδικασίας. Θέλουμε να έχουμε σχέσεις ε, που να δίνουν αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε εδώ και θα δώσω εδώ το λόγο στην πρόεδρο της Βουλγαρικής Βουλής, κυρία Καρατζέγεβα. Παρακαλώ. господин Αξιότιμε πρόεδρε, κύριε Ταγιάννη, κύριε Επίτροπε Ντομπρόφσκη, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Ως πρόεδρος ε, της Βουλγαρικής Εθνοσυνέλευση, θα ήθελα να εκφράσω την ε, ευχαρίστηση που νιώθω που μπορώ να συμπροεδρεύω αυτής ε, της κοινοβουλευτικής συνέλευσης για τη σταθερότητα και την οικονομική διακυβέρνηση και συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για την τρίτη σχετική εκδήλωση σε σχέση με την ε, διακοινοβουλευτική διάσταση που οργανώνει η Βουλγαρική Προεδρία και είναι η πρώτη εκδήλωση που λαμβάνει η χώρα εδώ στις Βρυξέλλες, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, οικοδεσπότες για τη φιλοξενία τους. Αυτό που μας φέρνει εδώ σήμερα όλους είναι η ανάγκη να συνεργαστούμε για να πετύχουμε την οικονομική σταθερότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι χαρά και τιμή μου που μπορώ να κηρύξω τις ενέργειες των εργασιών για το πρώτο κομμάτι της σημερινής αυτής ε, συνεδρίασης που έχει ως τίτλο την ενδυνάμωση της αντοχής και της σταθεροποίησης της ε, ΟΝΕ. Υπάρχει δηλώση της θα ήθελα να ζητήσω κι εγώ να επικρατήσει ενότητα σήμερα περισσότερο από ποτέ. Αυτή είναι άλλωστε ε, αυτό το σλόγγαν ε, που έχουμε και ως Βουλγαρική Προεδρία ισχύσεν τη ενώση. Ωστόσο αυτό το πολιτές μεσονομικό πλαίσιο Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θέλουμε να ενδυναμώσουμε την οικονομική διακυβέρνηση, να έχουμε ένα σημαντικό όραμα και πρέπει να προωθήσουμε κοινέ πολιτικές. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχρηματοδοτεί πολιτικές σε συγκεκριμένους ε, σημαντικούς τομείς της οικονομίας των κρατών μελών, ενισχύοντας την οικονομική, κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο. Πρέπει να είμαστε επίσης ευέλικτοι και αποτελεσματικοί. Έξω και θα ήθελα εδώ να δηλώσω ότι η Βουλγαρία στο εξάμεινο της Προεδρίας της εργάζεται για την περαιτέρω ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής ε, της ε, Νομισματικής και Οικονομικής ε, Ένωσης. Είναι μια προτεραιότητα, όπως είναι και η μεγαλύτερη δημοκρατική λογοδοσία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων απέναντι στους πολίτες που εκπροσωπούν. Γι' αυτό και χαίρομαι πολύ που εδώ συζητούμε μια νέα προσέγγιση και που κάνουμε συζητήσεις σε βάθος για το θέμα αυτό. Στο πλαίσιο αυτών των κοινών συζητήσεων θα δούμε ποιες είναι ευρωπαϊκές προοπτικές για ένα καλύτερο συντονισμό των ε, νομισματικών πολιτικών και των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών. Κάτι επίσης πολύ σημαντικό πρέπει να εστιάσουμε σε ζητήματα που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την Ευρωζώνη, για παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκομίσει όφελος εάν ενταχθούν στην Ευρωζώνη περισσότερα κράτη-μέλη. Το έχει πει ξεκάθαρα και ο πρόεδρος Γιούνκερ. Πρέπει να συζητήσουμε και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι κάτι που θα επηρεάσει αρνητικά και τον νοσιακό προϋπολογισμό. Το Brexit πρέπει να το συζητήσουμε γιατί θα επηρεάσει τη χρηματοδότηση των πολιτικών στο μέλλον. θα επηρεάσει και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε επιπτώσει θα τις δούμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία από τις προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας είναι να περιοριστούν οικονομικές ε, και κοινωνικές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών. Επιμένω λοιπόν ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να διατηρήσει τον προεξάρχοντα ρόλο της και στο μέλλον. Είναι μια πολιτική η οποία αφορά επενδύσεις στις εθνικές υποδομές, αφορά τις ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, την χρηστή διακυβέρνηση. Είναι μια άκρο σημαντική πολιτική για εμάς, αλλά και για όλους υποθέτω. Έξω και είναι προτεραιότητα για τη Βουλγαρική Προεδρία, όπως είπα, διότι πρέπει να γεφυρώσουμε τις διαφορές μας. Καλωσορίζω τις προσπάθειες και της βουλγαρικής κυβέρνησης αλλά και των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για περιορισμό των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα. Χαίρομαι που ακολουθούν ε, το μονοπάτι για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Θα πρέπει να δούμε και την Ένωση των Κεφαλαίων Αγορών, πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη αντοχή στο τραπεζικό σύστημα πρέπει να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να βελτιώσουμε την διάρθρωση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Εν κατακλείδη, το κλειδί για τη σταθεροποίηση και την ευημερία στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει να δράσουμε με υπευθυνότητα με ισορροπημένο τρόπο να είμαστε επικοδομητικοί και φιλόδοξοι. Έτσι θα πετύχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριο Βάλτης Ντομπρόφσκης, αρμόδιος για το χαρτοφυλάκιο για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο. Έχετε το λόγο. Αξιότιμοι κύριοι Πρόεδρε, Πρόεδροι, Ταγιάννη και Καραντσάγεβα, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας μιλήσω για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η συζήτηση αυτή τη στιγμή έχει επεκταθεί, είναι πολύ ζωντανή και έχουμε πει πολλά για τη μεταρρύθμιση της ΟΝΕ, κάτι το οποίο δεν θα είναι εύκολο. Επομένως, σε πολύ ε, επίκαιρο χρονικό σημείο έρχεται η διοργάνωση της εκδήλωσής σας. Οι οικονομικές προοπτικές είναι καλές. Είμαστε στην έκτη συνεχή χρονιά οικονομικής ανάπτυξης. Η ανάπτυξη έχει επιστρέψει σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα έχουμε ξεπεράσει τις προσδοκίες πέρσι και επιταχύνουμε το ρυθμό μας στην ανάπτυξη και στη ζώνη του ευρώ αλλά και εκτός ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ανάπτυξη θα είναι 2,7% το 2017 θα κλείσει τελικά το ταχύτερο της δεκαετίας και αυτή η ταχύς ρυθμής ανάπτυξης θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια όπου περιμένουμε ρυθμούς 2,9-2,1% αντιστοίχως. Άρα η οικονομία της Ευρώπης είναι εύρωστη, η ανεργία είναι στα χαμηλότερα επίπεδα της δεκαετίας, η ζήτηση είναι ισχυρή και η στήριξη των χρηματοπιστωτικών συνθήκων είναι ευνοϊκή για τις περισσότερες επενδύσεις και δημιουργία ευκαιριών για να προχωρήσουν όλοι προς τα εμπρός. Η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών είναι ισχυρή και αυτό θα οδηγήσει σε ακόμα καλύτερες οικονομικές επιδόσεις στο μέλλον. Βεβαίως υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι από τη στιγμή που η μεταβλητότητα των χρηματαγορών πρόσφατα μας δείχνει ότι ε, διαχειρίζεται τους κινδύνους και επιτυχάνεται σημείο ισορροπίας ε, βραχυπρόθεσμο. Πρέπει να επαναξιολογήσουμε τους κινδύνους. Παραμένει η πολιτική αβεβαιότητα λόγω των διαπραγματεύσεων για το Brexit και λόγω του κινδύνου ε, μεταστροφής, εσωστρέφειας σε προστατευτικές πολιτικές στο διεθνές τερέωμα. Βεβαίω οι προεπτικές είναι διαφορετικές από μία χώρα σε χώρα, γιατί κάποιες χώρες άρχισαν να ανακάπτουν πολύ νωρίτερα από κάποιες άλλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε υψηλό χρέο και υψηλή ανεργία σε ορισμένες χώρες μόνο. Σε γενικέ γραμμέ όμω, οι οικονομικέ προοπτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλέ και έχει έρθει η ώρα να δείξουμε ότι μπορούμε να δράσουμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτό κρίση. Έχουμε παρουσιάσει το όραμά μα για την ΟΝΕ στην έκθεση των πέντε προέδρων του 2015 αλλά και στην ανακοίνωση που δημοσιεύσαμε πέρσι για την εμβάθυνση της ΟΝΕ. Εκτεταμένες συζητήσεις έχουν γίνει και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο και θέλω να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω θερμά και τα Εθνικά Κοινοβούλια για τις προτάσεις, τις εισηγήσεις τους έχουν συμβάλει και εκτιμούμε ιδιαίτερο στη συμβολή τους. Το πακέτο, η δέσμη μέτρων που παρουσιάστηκε το Δεκέμβριο παρουσιάζει ένα οδικό χάρτη δράση για συγκεκριμένες προτάσεις με βάση τις πιο πιεστικές ανάγκες και την πρόσφατη συζήτηση που έχει γίνει. Τονίζουμε αυτή την ιδέα του οδικού χάρτη, του χάρτη πορείας, γιατί πρέπει να δρούμε και βραχυπρόθεσμα, αλλά να έχουμε και όραμα μακροπρόθεσμο συνάμα και να ξέρουμε προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί η ΟΝΕ και μετά το 2019 αλλά και μετά το 2025. Οι αρχές για την ε, Κομισιόν είναι σαφείς. Ενότητα, αποτελεσματικότητα και δημοκρατική λογοδοσία. Ενότητα διότι το μέλλον και των χωρών της ζώνης του ευρώ και των χωρών που δεν είναι στο ευρώ είναι συνδεδεμένο και όλες οι χώρες έχουν νομικώς δεσμευτεί κάποια στιγμή να, προχωρήσουν, να προσχωρήσουν στο ευρώ εκτός από τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Και άρα αυτό θα είναι ανοιχτό για όλα τα κρατημένα. Αποτελεσματικότητα. Η ΟΝΑ, η χρειάζεται καλύτερη χρήση των υφιστάμενων εργαλείων και πιο σωστούς κανόνες και δημοκρατική λογοδοσία, διαφάνεια για το ποιο αποφασίζει τι, μεγαλύτερος διάλογος με τους Ευρωπαίους εταίρους, με τα εθνικά κοινοβούλια, με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών με τους κοινωνικούς εταίρους. Όλα αυτά είναι απολύτως απαραίτητα. Υπάρχει μια χρονιά ολόκληρη, 12 μήνες νομοθεσίας, νομοθετικής δράσης πριν τις εκλογές, τις ευρωεκλογές και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία να προχωρήσουμε, να μην τη χάσουμε. Ο δικός χάρτης προβλέπει προτεραιότητα στην οριστικοποίηση της Τραπεζικής Ένωσης και καλωσορίζουμε την πολιτική βούληση και δέσμευση των ηγετών να ε, κάνουν τα απαραίτητα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Πρόοδο θα έχουμε μόνο εάν ε, ο στόχος για τη μείωση του ρίσκου και ο στόχος για το μοίρασμα των κινδύνων και των ρίσκων ε, συνοδεύει ο ένας τον άλλον και πάνε χέρι με χέρι έτσι ώστε και οι τράπεζες να παίξουν το ρόλο που τους αναλογεί και να χρηματοδοτήσουν την οικονομία, να μπορέσουν να δώσουν δάνεια για επενδύσεις για να παραμένουν οι επιχείρησεις ανταγωνιστικές. Πριν από ένα χρόνο παρουσιάσαμε ένα περιεκτικό πακέτο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών τραπεζών. Μαζί με τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό παρακολουθούμε εκ του σύνοικη στην υγεία του χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού κλάδου και πολύ προόδο έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με, τα, ε, με τις εκθέσεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα τελευταία τρία χρόνια το μερίδιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει μειωθεί κατά το 1 τρίτο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του 2017, ο λόγος είναι στο 4,6% των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως υπάρχουν τεράστιες διαφορές, μεγάλες διαφορές μεταξύ χωρών από τη μία χώρα στην άλλη και σημαντική είναι η πρόοδος και στα κράτη-μέλη που αρχικά είχαν πολύ μεγάλο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων και πολύ μεγάλο ποσοστό μη ε, ε, εισερχόμενων μεταρρυθμίσεων. Εκεί έχουμε μεγάλη πρόοδο. Και θα παρουσιάσουμε και άλλες προτάσεις για τη μείωση του βάρους των μη εξυπηρετούμενων δανείων και για την πρόληψη της ισόρευσης μη εξυπηρετούμενων δανείων στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα κοινό backstop για το Single Resolution Fund, για το κοινό Ταμείο Εξυγίασης των Τραπεζών και για το, ε, την ενιαία Ευρωπαϊκή Εγγύηση Καταθέσεων. Η ισχυρή προστασία των καταθέσεων, ακόμα και όταν μια κρίση χτυπά ένα κράτος μέλος, θα οδηγήσει να προστατεύσουμε το κράτος μέλος από μπάνκραν, από διαφυγή κεφαλαίων και από κινήσεις πανικού. Δεν θα πρέπει βεβαίως η ενιαία ευρωπαϊκή τραπεζική εγγύηση καταθέσεων να δημιουργεί ηθικό κίνδυνο, moral hazard. Θα πρέπει όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη και να τα προχωρήσουμε με σταδιακό τρόπο. Εξού και όλα αυτά είναι εργαλεία και για, το, και για τη μείωση του κινδύνου αλλά και για το μοίρασμα, το καλύτερο μοίρασμα των κινδύνων έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας θα το μετατρέψουμε σε Ευρωπαϊκό ε, Νομισματικό Ταμείο. Θα πρέπει να αγκιστρωθεί θεσμικά στα θεσμικά όργανα, να δημιουργηθούν συνέργειες και να υπάρχουν απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας για διαφάνεια και λογοδοσία. Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα είναι το backstop για το Single Resolution Fund, για το ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης Τραπεζών. Και θα Πιστεύουμε ότι υπάρχει στην αρχιτεκτονική αυτή τη στιγμή, στην αρχιτεκτονική δομή, ε, καλή ισορροπία και ε, θα πρέπει να παραμείνει ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων αρκετά ισχυρός. Δεύτερη πρωτοβολία είναι πρόταση να μπει στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η ουσία της συνθήκης για το συντονισμό ε, στην ΟΝΕ, δηλαδή το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Τα, οι χώρες που το υπέγραψαν είναι σε θέση να ολοκληρώσουν αυτή την πρόθεσή τους και να τους συμπεριλάβουν να γίνει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία κανονική όπως προβλέπεται και στις συνθήκες. Όλο αυτό θα απλουστεύσει το νομοθετικό πλαίσιο και θα κάνει να αποφύγουμε τις νομοθετικές επικαλύψεις. Θα ενισχύσει τη λογοδοσία και η πρόταση περιλαμβάνει τη διατήρηση του ρόλου των Εθνικών Κοινοβουλίων και των συζητήσεων όπως αυτές που γίνονται εδώ σήμερα. Στόχος είναι να ενισχυθούν οι εθνικές διαδικασίες για υγιή δημόσια οικονομικά. Η πρόταση της Κομισιόν δεν επηρεάζει το παράγωγο δίκαιο σε σχέση με τη σταθερότητα και το σύμφωνο ανάπτυξης. Θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε τα δημόσια οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ανταποκριθεί η Ένωση στις προκλήσεις. Πέρσι συμβάλαμε στη συζήτηση για την επόμενη σύνοδο για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020. Είχαμε προτάσει για το πώ θα τα δημόσια οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να στηρίξουν περισσότερο τις εθνικές επενδύσεις και να στηρίξουν τις χώρες. Θέλουμε να δώσουμε επιπρόσθετη στήριξη στα κράτη-μέλη και να τα βοηθήσουμε να εφαρμόσουν τις εθνικές μεταρρυθμίσεις όπως έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν προτάσεις και για την περίοδο μετά το 2020. Αυτή τη στήριξη τη δοκιμάζουμε και την έχουμε ήδη σήμερα το 2018 μέχρι 2020 με εθελούσια κινητοποίηση μέρος του αποθεματικού ε, των Ευρωπαϊκών Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων. Έχουμε πρόταση νομοθετικής τροπολογίας για το ε, κανονισμό που διέπει τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και κοντήλια. Θέλουμε για την περίοδο 2018 και 2020 προτείνουμε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του ε, προγράμματος στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ε, με πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από τα ήδη διαθέσιμα. Είναι ένα πρόγραμμα πολύ δημοφιλές από την έναρξή του. Με αυτό το πρόγραμμα στηρίζονται 150 έργα σε 15 κράτη-μέλη και είμαστε στη διαδικασία επιλογής νέων έργων για τη φετινή χρονιά. Για το 2018... Η ζήτηση προήλθε από 20 κράτη-μέλη και περισσότερα και ήταν πενταπλάσια από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Εξού και προτείνουμε την ενίσχυση και την αύξηση του προϋπολογισμού για να ανθίσει το ευρώ ακόμα περισσότερο και να ανθίσουν και οι χώρες εντός του ευρώ πρέπει να έχουμε σύγκληση. Πρέπει να έχουμε περισσότερη τεχνική στήριξη αναλόγως με τα αιτήματα της κάθε χώρας και να τη στοχεύσουμε στους κλάδους και στους τομείς που μπορούμε να πετύχουμε υψηλή σύγκληση. Δημόσια διαχείριση των οικονομικών, αγορά εργασίας, αγορά προϊόντων, ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης και ούτω καθεξής. Προτείνουμε να έχουμε δημοσιονομική σταθεροποίηση, ε, ένα ταμείο για τη δημοσιονομική σταθεροποίηση στις χώρες του ευρώ για να υπάρχει καλύτερη προστασία έναντι των ασύμετρων σοκ και μπορούμε να συμπληρώσουμε έτσι το ρόλο των εθνικών προϋπολογισμών. Οι επενδύσεις έρχονται πρώτα από τον εθνικό προϋπολογισμό σε χαλεπούς καιρούς και αυτό έχει αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και στην ανάπτυξη. Στήριξη μπορεί να έρθει από διάφορες πηγές χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δάνεια κατά κύριο λόγο και... Αυτές οι ιδέες θα γίνουν πολύ πιο συγκεκριμένες στην νομοθετική πρόταση που θα υποβάλουμε για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή η λειτουργία σταθεροποίησης θα ελαχιστοποιήσει τον εθνικό ε, κίνδυνο και θα υπάρχουν σαφή κριτήρια επιλεξιμότητας. Βεβαίως πρέπει τα κράτη-μέλη στους ε, ε, καλούς καιρούς των παχιών αγελάδων να συνεχίζουν να χτίζουν κεφαλαιακά μαξιλάρια σε σχέση με τη θέση του Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομικών είμαστε υπέρ και πιστεύουμε ότι θα ε, ε, βοηθήσει την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα έρθει σε αντίθεση με τις εθνικές αρμοδιότητες και θα είναι υπόλογος και θα λογοδοτεί και στα εθνικά κοινοβούλια. Στην έκθεσή μας δίνουμε έμφαση στη δημοκρατική νομιμότητα το, του συντονισμού της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής και της ΟΝΕ αυτή, αυτής καθεαυτές. Η εντατική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μέρος της δημοκρατικής λογοδοσίας. Η, η, ε, η, η διαλεκτική με τα εθνικά κοινοβούλια επίσης και τους ομολόγους μας σε εθνικό επίπεδο. Η, μια ολοκληρωμένη ΟΝΕ μπορεί να είναι μόνο δημοκρατική. Η εβδομάδα αυτή είναι μια εξαιρετική πλατφόρμα για να τελειοποιήσουμε τις λεπτομέρειες ε, και να ενισχύσουμε τη δημοκρατική διαδικασία. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βασιστούμε στην ενεργή σας στήριξη. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστούμε πολύ, Αντιπρόεδρε Ντομπρόφσκης. Θα πρέπει να φύγετε για το Eurogroup στις 10 και 4, γι' αυτό ξεκινούμε αυτή αμέσως την συζήτηση. Επτά ε, έχουν ζητήσει τον λόγο. Δύο λεπτά. Παρακαλώ. Ο κύριος Ερικ Βέρ από την Επιτροπή Οικονομικών Αποθέσεων της Γαλλικής Βουλής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βεβαίως πρέπει να επιδιώξουμε να προχωρήσουμε σε το άμεσο χρονικό διάστημα σε πολλά θέματα, αλλά από αυτά που ανέφερε ο Αντιπρόεδρο, κατά πρώτον πρέπει να κοιτάξουμε να ε, μετριάσουμε του κινδύνου για την Τραπεζική Ένωση σε πρώτη φάση και να κοιτάξουμε και την Ένωση των Κεφαλαγορών. Κατά δεύτερον, ο ευρωπαϊκό προπολογισμό είναι πολύ αδύναμο, πολύ περιοριστικό και αυστηρό. Βεβαίω πρέπει να γίνεται σεβαστή η ταυτότητα τη κάθε χώρα και υπάρχουν πολιτικέ που υλοποιούνται εδώ και πολύ καιρό, Όμω χρειαζόμαστε έναν ε, προπολογισμό πιο ενισχυμένο για να μπορούμε να παρέμβουμε. Και το τρίτο σημείο είναι ότι πρέπει να αποφύγουμε την φορολογική ε, διάθεση να μην γίνονται σεβαστοί κανόνε. Ε, Ιδίω στην ε, Ευρωζώνη πρέπει να υπάρχει κάποια φορολογική ένωση. Ε, Μα έχει ανησυχήσει πολύ το θέμα αυτό επίση και το πώ θα φορολογήσουμε τι ψηφιακέ συναλλαγέ. Ε, πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε να υπάρξουν πολιτικές αποφάσεις που να συνοδεύουν τις οικονομικές αποφάσεις. Το βλέπουμε διαρκώς ε, στα κοινοβούλια στις χώρες μας, αλλά ακόμη περισσότερο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι κάτι τέτοιο χρειάζεται. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ποιο είναι το πραγματικό χρονοδιάγραμμα, το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δώσει μια χειροπιαστή απάντηση σε αυτό το φαινόμενο που ε, μένει ε, και δεν μπορεί κανείς παρά να πει ότι είναι άδικο. η Γκάφα και όσοι ε, ε, οι εταιρείε αυτές και όσοι τις χρησιμοποιούν δεν πληρώνουν τους φόρους που πρέπει. Ο Τζαν Πάολο Γκάλι από την ε, Ιταλική Βουλή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο δικό μας κοινοβούλιο ήδη εγκρίναμε τον Δεκέμβριο Ε, το μεγαλύτερο μέρος ε, του προγράμματος εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018 και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τομπρόφσκης ε, για τα σημεία που ανέφερε σε συνδυασμό με την ομιλία του Πρόεδρου Ταγιάννη. Απλώς να κάνω μία παρατήρηση. Έχει γίνει μια σειρά από προτάσεις που κυκλοφορούν στην Ευρώπη, όχι αναγκαστικά από τους ανώτερους αξιωματούχους, για την ε, ε, αναδιάρθρωση των ε, δημόσιων χρεών. Αυτό από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, τον κύριο Σόιμπλε, και από σχετική του δήλωση, κάποιο κείμενο που κυκλοφόρησε και από Γερμανούς και Γάλλους οικονομολόγους πρόσφατα σε άλλο κείμενο, σε άλλο δημοσίευμα. Μήπως λοιπόν η ενίσχυση της ανθεκτικότητας, που είναι ο τίτλος αυτού του πάνελ, είναι κάτι που ε, δεν θα προσφέρει σταθεροποίηση στην Ευρωζώνη. Αυτή η αναδιάρθρωση ίσως να είναι σε κάποιες περιπτώσεις απαραίτητη, αλλά αν ορίσουμε και τους κανόνες κεντρικά, διατρέχουμε τον κίνδυνο να ε, πέσουμε σε μια αυτεκπληρούμενη προφητεία η αναδιάρθρωση μπορεί να λειτουργήσει αν είναι πια οριστική. Δηλαδή στο επόμενο βήμα η κυβέρνηση να μην χρειάζεται να ε, πηγαίνει στις αγορές για να καλύψει τις ανάγκες της. σε κάποιες χώρες το κούρεμα του χρέους κατά 50% θα δημιουργήσει μια τεράστια ύφεση όχι μόνο στην ίδια τη χώρα αλλά σε όλη την Ευρώπη. Ε, οπότε δεν θέλουμε αυτοεκπληρούμενες προφητείες. όπως έγινε στη λεγόμενη, στο λεγόμενο περίπατο της Ντοβίλ όταν ο Σαρκοζίκη Μέρκελ με τις συζητήσεις του τελικά φάνηκε να εντείνουν τα προβλήματα της Ευρωζώνης. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια γενής αντίφαση. Εάν κάποιοι Ευρωπαίοι θύνοντες, κάποιες εθνικές αρχές τις επόμενες εβδομάδες ή ημέρες κάνουν δηλώσεις για το χρέος, την ε, αυτόματη αναδιάρθρωση του χρέου ή ένα σχετικό κανόνα, σε Ευρώπη διατρέχει τον κίνδυνο να αποσταθεροποιηθεί σοβαρά. Δεν ξέρω αν θα συμβεί κάτι ανάλογο με αυτό που έγινε μετά την ε, περίπτωση του Ντοβίλ. Αλλά διατρέχουμε αυτό τον κίνδυνο. Ευχαριστούμε κύριο Παπαδημούλη, Αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε τώρα που τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα για την ευρωπαϊκή οικονομία, αντιπρόεδρε Ντομπρόφσκης, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε τα βήματα μεγαλύτερης ευάθυσης και ενοποίησης της ένωσης που έχουμε. Γιατί έχουμε μια ατελή οικονομική ένωση, μια ατελή νομισματική ένωση και μια ατελή τραπεζική ένωση. Και πρέπει να προετοιμαστούμε ενισχύοντας τις ενώσεις αυτές, θωρακίζοντάς τες, ολοκληρώνοντάς τες απέναντι στην κρίση που έρχεται. Τώρα που όπως είπε ο πρόεδρος Γιούνκερ δεν βρέχει, τώρα είναι η ευκαιρία να φτιάξουμε τη στέγη, γιατί αργότερα θα είναι πολύ αργά. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε και τη φορολογική εναρμόνιση. Βλέπετε τις αποκαλύψεις από τα σκάνδαλα. Panama Papers, Paradise Papers, δημοσιογράφοι ανακαλύπτουν σκάνδαλα που δεν μπορούν να ανακαλύψουν και να αποφύγουν οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί και οι κρατικοί προϋπολογισμοί και χάνουμε δισεκατομμύρια ευρώ και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτήν την τεράστια φορολογική απάτη των υπερπλουσίων που είναι νόμιμη ή νομιμοφανής αλλά είναι εξαιρετικά άδικη και ανήθικη. Και πρέπει απέναντι σε αυτό να κάνουμε βήματα φορολογικής αναρμόνισης. Δεν μπορούμε να έχουμε ο καθένας το δικό του φορολογικό σύστημα με μαύρες τρύπε σε βάρος των άλλων. Και το τρίτο, είναι αδύνατο να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερα πράγματα με λιγότερα χρήματα. Διότι στα τελευταία χρόνια έχουν προσθεθεί καινούριες προκλήσεις. Το προσφυγικό, το μεταναστευτικό, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η πίεση να κάνουμε περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει, αν θέλουμε και συμφωνώ με την πρόεδρο της Βουλγαρικής Βουλής, να προστατεύσουμε την πολιτική συνοχής, πρώτον ολοκληρώνω κύριε πρόεδρε οι χώρες που ωφελούνται περισσότερο από την ένωση και είναι οι πλουσιότερες όπως η γερμανία και η ολλανδία να δώσουν περισσότερα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και δεύτερον να αποκτήσουμε και ίδιους πόρους περισσότερου, περισσότερους αξιοποιώντας τις προτάσεις της Επιτροπής Μόντι. Σας ευχαριστώ από τη Δανέζικη Βουλή, ο εκπρόσωπός της και μετά ο αντιπρόεδρος Ντομπρόφσκης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ και να ξεκινήσω λέγοντας κάτι διαφορετικό. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το να ενώνει κανεί 27 χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δείγμα δημοκρατία στην Ευρώπη, ειρήνη και προόδου. Όμω ανησυχώ όταν χώρε θέλουν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν υπάρχουν αντιρρησίες όταν υπάρχουν διαφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανησυχώ για το εγχείρημά μας, διότι πιστεύω στην ειρήνη και τη δημοκρατία που μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ανησυχώ για τις χώρες που προσπαθούν να οπισθοχωρήσουν, να επαναχωρήσουν σε κάποιες από τις θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κοιτάξει αυτές τις περιπτώσεις και να προσπαθήσει αυτές τις χώρες να προχωρήσουν. Αυτά τα φαινόμενα να μην συμβαίνουν, να μπορούν ε, οι πολίτες να ενδιαφέρονται γνήσια για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δουλεύουν για αυτήν. Ε, ε, σε σχέση με όσα λέμε τώρα όμως, νομίζω ότι είναι πολύ θετικό αυτό που υπόθηκε για τι μεταρρυθμίσει. Στην Δανία κάναμε πολλέ μεταρρυθμίσει τα τελευταία 15 χρόνια. Έχουμε ορίσει διαφορετικά την ηλικία συνταξιδότηση, έχουμε κάνει την αγορά εργασία πιο ευέλικτη και αυτό για να έχουμε καλύτερα, ε, καλύτερη οικονομία σε κρατικό επίπεδο να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές ανάγκες. Νομίζουμε ότι όλες οι χώρες πρέπει να κοιτάξουν ε, εσωτερικά τις ε, οικονομικές τους υποθέσεις για να στηρίξουν λίγο την ε, οικονομία τους. Είναι μια εθνική, ένα εθνικό καθήκον αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνδράμει. Επίσης, τα θέματα των ανισοτήτων στη Δανία προσπαθούμε να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις ανισότητες, ακόμα και γεωγραφικώς. Νομίζω λοιπόν ότι από την άποψη των εθνικών μας καθηκόντων είναι σημαντικό και βεβαίω οι καλές ιδέες είναι κάτι που μπορεί να μας ε, βοηθήσει σε κάθε περίπτωση, αλλά νομίζω ότι πρέπει ο καθένα να βλέπει τα πράγματα και σε επίπεδο χώρα ε, και να αναλαμβάνει τι εθνικέ του Ο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε αξιότιμοι βουλευτές. Πρώτα απ' όλα, θέλω να ευχαριστήσω την υποστήριξη που εκφράσατε στο έργο μας για την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλογρών και της Τραπεζικής Ένωσης ως προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύω ότι σύντομα θα δούμε απτά αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα για το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων σε ό,τι αφορά την εμβάθυνση της ΟΝΕ. Υπάρχουν σημαντικά χρονικά σημεία όπως είναι η διάσκεψη κορυφής ε, του Μαρτίου αλλά και του Ιωνίου που ήδη ελπίζουμε να καταλήξουμε σε κάποιες ε, συμφωνίες σε ό,τι αυτό το πακέτο του Δεκεμβρίου για την εμβάθυνση της ΟΝΕ και τέλος το Μάιο του 2019 θα έχουμε ένα, μια επίσης ε, διάσκεψη κορυφής όπου ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα για το μέλλον της Ευρώπης στο πλαίσιο αυτής της κοινοβουλευτικής ε, περίοδου. Άρα έχουμε μπροστά μας πολύ σημαντικούς μήνες. Ετέθησαν πολλά ερωτήματα για τις προτεραιότητες του ενωσιακού προϋπολογισμού, για το μέγεθος του ενωσιακού προϋπολογισμού και πράγματι, όπως γνωρίζετε, πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε τη δική της πρόταση στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής για το προσεχές ε, πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Και εμείς ε, είμαστε της άποψης ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρές ε, προκλήσεις ε, με το Brexit ε, ανοίγει μια μεγάλη τρύπα στον προπολογισμό. Άρα σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι κάτω του 1% ε, σε σχέση με το ΑΕΠ ο ενωσιακός προπολογισμός, αλλά πολύ περισσότερο. Πρέπει λοιπόν να καλύψουμε την τρύπα του Brexit, αλλά και να μπορέσουμε να καλύψουμε τις νέες προτεραιότητες. Γι' αυτό θα χρειαστεί επανειεράρχηση των προτεραιοτήτων σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, αλλά θα πρέπει να μεγαλώσει και ο νοσιακός προπολογισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν εργάζεται και προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις και σε ό,τι αφορά τους ίδιους πόρους επίσης πρόθεσή μας είναι να καταθέσουμε τις προτάσεις μας για ενδεχόμενους νέους ίδιους πόρους. Ετέφθη ένα ερώτημα για την αυτόματη αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους. Αν δείτε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα δείτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτείνει έναν τέτοιο μηχανισμό. Φυσικά και αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση και θεωρούμε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτή τη συζήτηση για να μην υπονομεύσουμε την ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να έχουμε υπόψη και ενδεχόμενες αρνητικές ε, συνέπειες. Στόχος είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΩΝΕ, όπως και ε, τονίσαμε προηγουμένως. Επίσης αναφέρθηκε το θέμα της φορολογίας από αρκετούς ομιλητές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά και συμφωνεί πλήρω. Σε ό,τι αφορά την φορολογία, πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν. Και έχουμε ήδη επιτύχει σημαντική πρόοδο τα δύο-τρία τελευταία έτη. Τροποποιήσαμε την οδηγία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής φοροαποφυγής. Έχουμε συνάψει συμφωνίες για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μέλων για την πάταξη της φοροαποφυγής, αλλά έχουμε και συμφωνίες με τρίτες χώρες. Υλοποιήθηκε επίση η πρωτοβουλία του ΟΣΑ κατά τις μετατόπιση κερδών διάβρωση βάση και έχουμε και ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων για το ΦΠΑ και την καταπολέμηση του διεθνούς ε, της ε, φοροδιαφυγής ε, σε ό,τι το διεθνή ΦΠΑ. Έχουμε τις εκθέσεις αναχώρα, τις προτάσεις μας για την κοινή ενιαία ε, βάση φορολόγησης επτεριών. Θα έχουμε και τις προτάσεις μας σύντομα για την ψηφιακή φορολογία, για να μπούμε δυναμικά στην ψηφιακή εποχή. Άρα στον τομέα της φορολογίας ήδη έχουμε ένα θεματολόγιο σημαντικό και η αρχή που μας διέπει είναι να φορολογείται το κέρδος εκεί που γίνεται η οικονομική δραστηριότητα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις παρατηρήσεις και τα σχόλια σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του ρόλου και των κρατών μελών και των εθνικών κοινοβουλίων και εθνικών κυβερνήσεων σε ό,τι αφορά τη χάραξη οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής που να είναι σοβαρή και αποτελεσματική. Μπορούμε να ενισχύσουμε εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά αυτά τα εργαλεία δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση σε εθνικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ντομπρόφσκης, για την, για παρουσία σας. Πριν το διάλειμμα, η κυρία αγόρτες, θα λέμε το λόγο, κυρία Σπέτσα από την Κροατία. Ευχαριστώ ε, για την πρόσκληση. Για την Κροατία, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, που δεν είναι ακόμη μέλος της Ευρωζώνης, είναι πολύ σημαντική. Όπως ακούσαμε ήδη από τις διάφορες ομιλίες του Ευρωκοινοβούλιο, ε, η Ευρωζώνη μπορεί να προσφέρει ωφέλη, και αυτό είναι στρατηγικό στόχο για μας. Η Κρατική Βουλή και η Τράπεζα τη Κροατία έχουν παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ε, με σκοπό την προσχώρηση στο ευρώ που έχει γίνει αντικείμενο δημόσιων συζητήσεων στη χώρα. Θέλουμε να γίνουν γνωστά τα ωφέλη της προσχώρησης στην Ευρωζώνη σε όλους τους πολίτες της Κροατίας. Είμαστε μια χώρα που πληρώνουμε όλες τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχουμε στην Ευρωζώνη. Γι' αυτό μας ενδιαφέρουν όλες οι προτάσεις ε, από τη δεσμή μέτρων για την εμπάθυνση της ΟΝΕ. Ναι. Και μας ενδιαφέρει η αύξηση των κονδυλίων για την ενίσχυση των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν ακριβώς τις μεταρρυθμίσει και να φτάσουν να εκπληρώνουν τα κριτήρια για προσχώρηση στην Ευρωζώνη. Επίσης, καλωσορίζουμε το εργαλείο για την ε, ε, υλοποίηση των διευθυντικών αλλαγών. Τον Ιούνιο του 2017 βγήκαμε από τη διαδικασία του υπερβολικού ε, ελλείμματος και τώρα είμαστε σε πορεία σύγκληση με την Ευρωζώνη και ε, εξάλληψη των μακροοικονομικών ανισοτήτων. Είμαστε σε πιλωτικό στάδιο και θα παραμείνουμε σε αυτό έως το 2020 με το νέο μηχανισμό στήριξης που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν τα αποθεματικά του μηχανισμού. Το 2020 όλα αυτά θα εντάσσονται στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που τώρα ε, είναι ξεχωριστό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πάβελ Αριμάκη από τη Φιλανδική Βουλή. Παρακαλώ. το μικρόφωνο σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος Ταγιάννη έθεσε ένα θέμα, την ε, εμπιστοσύνη και την πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια, κατά τη διάρκεια της ε, κρίσης, είδαμε ότι η εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, περιορίστηκε. Βεβαίως, όταν ε, ο κόσμος, οι πολίτες πλήττονται από τις περικοπές στα κρατικά ε, δημοσιονομικά, υποφέρουν. Πρέπει λοιπόν αυτά τα θέματα να αντιμετωπίσουμε και να δούμε ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να τονώσει την απασχόληση, τις επενδύσεις που έχουν σκοπό τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, μπορεί να κάνει εδώ πολλά. Χρειαζόμαστε μια άλλη οπτική γωνία εδώ και πολλοί στην κοινωνία μας έχουν ε, πια την ε, αντίληψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για περικοπές που έχουν πλήξει τα πιο αδύναμα κομμάτια του πληθυσμού. Ότι οι θεσμοί της είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Ας δούμε όμως παραδείγματα όπως της Φιλανδίας. 3% μειώθηκε ο μισθός των βουλευτών στη χώρα μας, τη στιγμή που υπέφεραν ε, όμως πολύ περισσότερο νέοι και αδύναμα ακόμα και του πληθυσμού. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε περιπτώσεις που έχουν πλήξει την αξιοπιστία μας. Περιπτώσεις όπως ε, το σκάνδαλο LuxLeaks ή τα έγγραφα του Παναμά, Όλα αυτά επηρεάζουν τους φορολογουμένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παραμένουν ανενόχλητοι κάποιοι φορολογικοί παράδεισοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να κοιτάξει τι θα γίνει με τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, με τα συνταξιδοτικά. Δεν μπορούμε διαρκώς να έχουμε μια πορεία ε, ύφεση σε αυτά. Πρέπει, Αντιπρόεδρε Ντομπρόφσκης, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το φορολογικό dumping στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εντός των συνόρων πριν περάσουμε σε φορολογική ένωση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ταϊκούρας. with Βουλή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλο κόστος και πολλές δυσκολίες η Ευρωπαϊκή Ένωση σιγά σιγά εξέρχεται από την κρίση. Παραμένει όμως υψηλή αναργία, δημογραφικό πρόβλημα, προσφυγική κρίση, θέματα εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, Brexit, δημοσιονομική σταθερότητα, κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής. Η συλλογική απάντηση πρέπει να είναι μια πιο αθεκτική, ποιοτική Ευρώπη, ανταγωνιστική, αποτελεσματική, με ενισχυμένη αλληλεγγύη, εμβαθύνοντας και ενισχύοντας την ΟΝΕ να έχουμε καλύτερο οικονομικό συντονισμό, επαρκή εργαλεία και πόρους για να αντιμετωπίσουμε τις ανισορροπίες. Συγκεκριμένα εργαλεία για μακροπρόθεσμη οικονομική διακυβέρνηση. Χρειαζόμαστε εφαρμογή υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών, πράγματι λαμβάνοντας, που θα λαμβάνουν υπόψη τον οικονομικό κύκλο. Πρέπει να υιοθετήσουμε ρεαλιστικούς δημοσιονομικούς στόχους και βελτίωση των δημοσίων οικονομικών με μείωση του βάρους της φορολογίας και καλύτερο έλεγχο των δαπανών, αντίθετα με αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Εφαρμογή συνεκτικών μόνιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, να οριστικοποιήσουμε να τελειοποιήσουμε την Τραπεζική Ένωση και να προχωρήσουμε σε μια πλήρη κεφαλαιακή ένωση που θα ανθίσει και θα ενισχύσει τη ρευστότητα. Και το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας πράγματι πρέπει να μετατραπεί σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, ένα εργαλείο σταθεροποίησης, δυνατότητα δανεισμού και δυνατότητα ανάπτυξης νέων οικονομικών εργαλείων. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κρέτσου από την Ρουμανική Βουλή. Καλό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ε, κυρίε και κύριοι, δεν έχουμε ακόμη ένα νόμισμα. Έχουμε ένα κοινό νόμισμα σε έναν ευρύτερο χώρο που ε, λειτουργεί σαν ε, ε με ξυλαράκι για να απορροφά του κρατασμού κατά μελών. Αυτό το νόμισμα θα μπορούσε όμως να λειτουργεί αποτελεσματικά ε, εάν μπορούσαν να εφαρμοστούν πολιτικές σύγκλησει για να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες. Βλέπουμε να αλλάζει κάπω το μοντέλο όμως από την αλληλεγγύη προς την κρατική ευθύνη. Και η κρατική υπευθυνότητα δεν μπορεί να ξεπεράσει τις ίδιες δυνατότητές της να παρέμβει και να ελέγξει τα αποτελέσματα με δημοσιονομικά εργαλεία για παρέμβαση. Τα κράτη-μέλη ήδη έχουν μεταφέρει και μοιραστεί ε, ε, αρμοδιότητες. Χρειάζονται λοιπόν πλέον ευρωπαϊκά εργαλεία παρέμβασης, εργαλεία αλληλεγγύης που για την ώρα δεν έχουμε. Η, ε, ανάληψη κοινών ε, κινδύνων εντός της εσωτερικής αγοράς δεν υπάρχει ελπίζω ότι ε, δεν θα ισχύσει αυτό που λέει μια ομάδα οικονομολόγων και να μην συμβουλεύουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μόνο ε, τα ανώτερα κλιμάκια των μάνατζερ θα γλιτώνουν την οικονομική κρίση. Αυτή τη στιγμή τιμωρούνται κράτη-μέλη με δημοσιονομική πειθαρχία, με πλήγματα στη δημόσια διοίκηση και το δημόσιο τομέα και με άειλα κέρδη, κέρδη που κανείς ε, δεν μπορεί να λάβει τα ωφέλη τους. Τα κράτη-μέλη όμως προσπαθούν να σεβαστούν τα κριτήρια αυτά και τελικά αυτοί που πλήττονται περισσότερο είναι οι καλοί μαθητές ε, όπως οι Ισπανοί και οι Ιρλανδοί φίλοι που θα μπορούσαν ε, να προσφέρουν τη μαρτυρία τους. Χρειάζονται λοιπόν αυστηρά κριτήρια αλλά δεν είναι αυτός ο τρόπος να ξεφύγουμε από την κρίση. Έχουμε αποδείξεις ότι έχουν εφαρμοστεί λανθασμένες πολιτικές. Το ισοζύγιο πληρωμών είναι πιο ε, σημαντικό, ιδίω εφόσον το πλεόνασμα του ενός μπορεί να είναι το έλλειμμα του άλλου. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και στον ιδιωτικό τομέα, στο υψηλό επίπεδο χρέωσης που υπάρχει εκεί, γιατί μπορεί να χρειάζεται και αναδιάρθρωση και των ιδιωτικών επενδύσεων. όπως συνέβη και στο παρελθόν. The last speaker... Ευχαριστούμε. Τελευταίος πριν από το διάλειμμα για καφέ, ο κύριος Κόπεσεκ από την Δημοκρατία της, της Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για να ενδυναμώσουμε την Ευρωζώνη και να υπάρξει σταθερότητα. Ανησυχώ όμως ότι κάποιες από τις προτάσεις που υπάρχουν θα αυξήσουν ε, το άγχος σε σχέση με την Ευρωζώνη. Βλέπουμε να έχει χωριστεί σε δύο ομάδες η Ευρωζώνη. Κάποιες είναι εύρωστες οικονομικά και κάποιες άλλες είναι αδύναμες. Όταν αντιμετωπίσαμε κραδασμούς και προβλήματα έπρεπε οι χώρες που είναι πιο δυνατές να βοηθήσουν τις πιο δύναμες. Εδώ είδαμε την πρώτη περίπτωση ε, ηθικού κινδύνου, θα έλεγα, που ε, έχει πλήξει την Ευρωζώνη. Επίσης, ως προς τις τράπεζες πρέπει να κοιτάξουμε τι θέλουμε να δημιουργήσουμε με τις τράπεζες που θα αναλαμβάνουν από κοινού τον κίνδυνο. Οι καταθέσεις των πολιτών μπορεί να ε, κινδυνεύσουν από ανάγκες πολιτών άλλων χωρών που δεν έχουν στα δημοσιονομικά. Για κάποιε χώρε λοιπόν μπορεί να προκύψουν προβλήματα στη δημοκρατία τη Τσεχία. Το τραπεζικό σύστημα είναι υγιέστατο και ανθεκτικότατο. Χρειαστήκαμε διάρθρωση, αλλά η εξυγίανση αυτή ήταν κάτι που ανέλαβαν οι Τσέχοι πολίτε. Τα προβλήματά μα τα λύσαμε μόνοι μα. Είμαι βέβαιο ότι διαφορετικά προβλήματα θα έχουν διαφορετικέ επιπτώσει στην κάθε χώρα. Άρα, μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων δεν είναι αναγκαστικά μονόδρομος. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχει διαφορετικό επίπεδο ολοκλήρωση σε διαφορετικέ χώρε τώρα ω προ την φορολογική εναρμόνιση. Δεν βρίσκω ότι είναι καλή ιδέα αυτή. Διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε θα υπάρχουν χώρε που θα προσπαθούν να έχουν χαμηλότερους φόρους. Ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίσουν να υπάρχουν χώρες που θα κάνουν την ανακατανομή τους μέσω του φορολογικού συστήματος με υψηλότερους φόρους. Τα πάντα θα εξαρτηθούν από την επιλογή του κάθε κάτους μέλους. Εν γέννη, η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να επιτρέψει περισσότερη ανάπτυξη. Δεν να προσπαθούμε κεντρικώ να τα ρυθμίσουμε όλα. Ε, τα Γιάννη, ευχαριστώ. Οι υπόλοιποι αγορητέ που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο θα μπορέσουν να λάβουν το λόγο μετά το διάλειμμα. Τώρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα για καφέ και θα συνεχίσουμε στι 11 ακριβώ. Εδώ στο ημικύκλιο με συζήτηση για το ρόλο των ε, κοινοβουλίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπότιτλοι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 σε το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 πρότεινα να

Gentlemen, please be so kind to take. Παρακαλώ καθίστε. Coffee break is always the most important. Το διάλειμμα για καφέ είναι πάντοτε το σημαντικότερο σημείο της μερίσιας διάταξης, γιατί επιτρέπει τη διαδικτύωση. Πάντως τώρα πρέπει να επανέλθουμε στις τακτικές εργασίες μας. Θέλω να σας καλωσορίσω, να καλωσορίσω όλους τους συμμετέχοντες από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θέλω να καλωσορίσω και τους Ευρωβουλευτές και αν με επιτρέπετε θα μιλήσω από εδώ και πέρα στη μητρική μου γλώσσα τα πολωνικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, η σημερινή Συνεδρίου ολομέλεια ε, θα έχει ως θέμα τον μηχανισμό σταθερότητας. Εργαζόμαστε όλοι σε σχέση με αυτόν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και από το Συμβούλιο και από την Κομισιόν για να προωθήσουμε τη σταθερότητα του συστήματος και να βελτιώσουμε τις αναπτυξιακές προοπτικές ε, της Ευρώπης. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να συζητήσουμε με ποιους τρόπους τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να συνεισφέρουν στη διαδικασία αυτή. και πώς μπορούν όλα αυτά που συζητούμε εδώ να μεταφραστούν ε, σε εθνικές λύσεις. Χρειάζεται σίγουρα και μια κοινή συνεννόηση και κατανόηση. Γι' αυτό λοιπόν θελήσαμε η σημερινή συζήτηση να έχει ως επίκεντρο, όπως είπα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Φυσικά θα μιλήσουμε και για την ε, Οικονομική και Νομισματική Ένωση, τον ε, Μηχανισμό Σταθερότητας και πώς αυτός ε, εφαρμόζεται και κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και κατά το Εθνικό. Χρειάζεται και η δική σας συμμετοχή χρειάζεται κι εσείς να περάσετε αυτό το μήνυμα στους πολίτες των χωρών σας. Αυτός είναι ο ρόλος μας ως Ευρωβουλευτών και Εθνικών Βουλευτών. Να επικοινωνούμε με τους πολίτες. Έχουμε λίγο πολύ μια μισή ώρα στη διάθεσή μας. Πώς θα οργανωθεί αυτή η συζήτηση. Θέλαμε όσο το δυνατόν περισσότεροι εξημών να λάβετε το λόγο. Να έχετε τη δυνατότητα να εκφράσετε τις απόψεις. Βέβαια δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος μας, οπότε αν θέλουμε να λάβουν το λόγο στο θετόν περισσότεροι, θα σας παρακαλέσω όλους να σεβαστείτε το χρόνο αγόρευσης που θα είναι δύο λεπτά, το πολύ τρία. Θα ακούσουμε δύο εθνικούς βουλευτές και έναν ευρωβουλευτή σε κάθε γύρο. Θα βλέπετε και το χρόνο, θα βλέπετε το χρονόμετρο και έχω και στο δεξί μου χέρι ένα εργαλείο, το βλέπετε, το σφυράκι μου, που θα χρησιμοποιήσω σε περίπτωση ανάγκης για να σας επαναφέρω στην τάξη. Η κυρία Στογιάνοβα η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Προπολογισμού τη Βουλγαρικής Εθνοσυνέλευση εκπροσωπεί τα Εθνικά Κοινοβούλια, συμπροεδρεύει μαζί μου, εγώ εκπροσωπώ Όπω καταλάβετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ακούσουμε και κάποιε εισαγωγικέ παρεμβάσει από γνωστού εσά. Ο πρώτο είναι ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη. Α ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα ήθελα καταρχά να δώσω το λόγο στην συμπρόεδρό μου, την κυρία Στογιάνοβα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λιμπεράτσκι, Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης και για το ότι προεδρεύετε και μας υποδέχεστε εδώ. Αξιότιμοι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, η Βουλγαρία είναι τώρα 11 χρόνια μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και έχω να πω ότι μετά από 11 χρόνια ξεκινάει και η Βουλγαρική Προεδρία, αυτό το εξάμεινο. Θέλουμε να δουλέψουμε για την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μια πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση, για μια ε, πιο ολοκληρωμένη οικονομική και νομισματική ένωση με περισσότερο βάθος, χωρίς να είναι όλα αυτά εις βάρος των ε, κρατών μελών που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Ε, είναι τιμή για μένα να συμπροεδρεύω στη σημερινή συνεδρίαση, η οποία θα ασχοληθεί με την περίοδο, μεταφορα... με την περίοδο τη μεταβατική, τη μετάβαση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας προς ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων σε αυτή τη διαδικασία. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ήταν πολύ σημαντικός κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης γιατί έδωσε επιπρόσθετη οικονομική στήριξη στα μέλη της Ευρωζώνης που αντιμετώπιζαν προβλήματα. Και τώρα λοιπόν αυτός ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας σιγά σιγά θα μετατραπεί, θα μεταμορφωθεί και θα πάρει τη μορφή ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Είναι κάτι που επιθυμούμε και διότι φρονούμε ότι θα πρέπει και τα κράτη-μέλη εκτός Ευρωζώνης να συνεργάζονται με αυτό τον μηχανισμό και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες της Ευρωζώνης, Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, λοιπόν, όταν δημιουργηθεί, να έχει την απαραίτητη την ικανότητα δανεισμού. Και γι' αυτό μιλούμε για τη θεσμική κατοχήρωση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, και γι' αυτό ε, λέμε ε, για την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων κατά την ε, εξέταση της λειτουργίας αυτού του μηχανισμού που θα γίνει νομισματικό ταμείο. Πρέπει λοιπόν τα εθνικά κοινοβούλια να έχουν τη δυνατότητα να αντιδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην επικουρικότητα και στην αναλογικότητα. Θα ήθελα να σας καλέσω να υποβάλλετε γενικότερα σχόλια για το ζήτημα αυτό, διότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για το μέλλον της Ευρώπης στο σύνολό της. Πρέπει όλοι να έχουμε υπόψη μας ότι θα διατυπώσετε τα σχόλιά σας, θα τα ακούσουμε ε, να μην μακρηγορείτε, να ακούσουμε πρώτα τους ομιλητές που βρίσκονται εδώ στο πάνελ. Ο, ο κύριος Γκουαλτιέρη είναι ο πρώτος που θα κάνει εισαγωγικέ παρατηρήσεις πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αναντήρητα ενισχυμένη δυνατότητα διαχείρισης θα είναι η βασική ραχοκοκαλιά της ε, ενισχυμένης ΟΝΕ. Γι' αυτό καλωσορίζουμε την πρόταση κανονισμού από το Συμβούλιο, του Συμβουλίου μάλλον, για την δημιουργία νέου κανονισμού, νέου μηχανισμού σταθερότητας. Όμως για την ώρα κάποιοι, ε, κάποια από όσα προτείνονται φαίνονται παραπλανητικά, διότι δεν έχουν να κάνουν με την ομισματική πολιτική που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ούτε ε, προς, ε, ερχόμαστε πιο κοντά στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να διατηρηθούν οι λειτουργίες ε, της μακρονομικής σταθεροποίησης που έχει τώρα ο ESM, καθώς και να ασχοληθεί με την, ανα, την ανακεφαλοποίηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εφόσον χρειαστεί δεν αλλάζουν πολλά πέραν από το όνομα ουσιαστικά από τον μηχανισμό σταθερότητα. Είναι βέβαια μεγάλη αλλαγή και αυτή, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να εισάγει κάποιε στοχευμένε βελτιώσει ε, στου κανόνε ε, για τον μηχανισμό, διατηρώντα τι τωρινέ αρμοδιότητε τη Επιτροπή στο πλαίσιο του ε, ευρωπαϊκού συντονισμού και τη μακροοικονομική επιτήρηση. Αυτό είναι μεν καλό γιατί η επικάλυψη αρμοδιοτήτων δεν θα ήταν μόνο παράνομη βάση των συνθήκων αλλά και αντιπαραγωγική ω προ τη μακροοικονομική συνέπεια. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε να μην αναθέσουμε την αρμοδιότητα στο νέο κανονισμό να ασχοληθεί με τη μακροοικονομική ανάλυση που αυτή τη στιγμή ε, γίνονται βάσει του άρθρου 4 Γι' αυτό θα πρέπει η αναδιάρθρωση του χρέους να είναι μια προϋπόθεση για την στήριξη του ESM, κάτι που για την ώρα έχει αποκλειστεί. Διότι αυτό θα έπληκε τη μικροκρομική σταθερότητα και θα ερχόταν σε αντίφαση με το ίδιο το καθήκον του ESM, όπως ορίζεται στο άρθρο 3.6 της συνθήκης. Εδώ λοιπόν διαβάζουμε κάποιες προτάσεις ε, των ε, πανεπιστημιακών που μπορεί να είναι εύστοχες, όμως εδώ η πολιτική και η υπεύθυνοι τη Κεντρική Τράπεζα φαίνεται να γνωρίζουν καλύτερα τα τη μικροοικονομική σταθερότητα που έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα. Εδώ καλωσορίζω την ε, ε, απόφαση του Γάλλου Υπουργού Οικονομικών. Κόκκινη γραμμή δεν θα συμβεί αυτό και είναι συνετό. Ένα βασικό στοιχείο όμω το οποίο θέλω να επικεντρωθώ ε, στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η συμπερίληψη στο νέο ESM, στο νέο ε, νομικό πλαίσιο βάσει του άρθρου 353 από τη Συνθήκη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι καθοριστική σημασία γιατί θα ενισχύσει την θεσμική συνέπεια και την ε, ε, συνοχή του δημοσιονομικού μας πλαισίου και θα δοθεί δυνατότητα να αποδοθούν επιπλέον αρμοδιότητες στον ESM από τη στιγμή που θα ενσωματωθεί στην Ένωση. Ένα παράδειγμα. Εφόσον ενσωματωθεί στις συνθήκες του ESM θα είναι πιο απλό να προσφέρει μακροοικονομική σταθερότητα στον ευρωπαϊκό προπολογισμό δίνοντας ένα backstop από την προοπτική του Κοινοβουλίου και για να φτάσουμε στο θέμα ε, που μας απασχολεί, πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είναι πια η διακυβερνητική μέθοδος αυτή που προτείνεται, αλλά μια διαδικασία του άρθρου 300, του 352, δηλαδή η ομοφωνία απαιτείται ακόμη σε επίπεδο κρατών μελών, ενώ στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων θα υπάρχει πλέον συμμετοχή και θα απαιτείται η διαφάνεια και η δημοκρατική λογοδοσία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Τα άρθρα 5 και 6 από την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπουν διατάξει για να υπάρχει ακριβώ αυτή η δημοκρατική λογοδοσία, βάσει τη οποία ο ESM και το IMF θα υποβάλλουν ετήσια έκθεση προ το Ευρωκοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και επίση προ τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωκοινοβούλιο καθώς και τα Εθνικά Κοινοβούλια μπορεί να ζητήσουν γραπτές απαντήσεις σε ερωτήσεις τους και να καλήσουν τον εκτελεστικό διευθυντή να τους μιλήσει. Η ρήτρα ευελιξίας είναι κάτι το οποίο θα τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν με την ομοφωνία του Συμβουλίου και τη συνένεση του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν όμως κάποια στοιχεία που του αφήνουν να υπονοήσουν ότι θα υπάρξει μια διελκυστίνδα εξουσίας μεταξύ αυτών και του Ευρωκοινοβουλίου για να πάνε πέρα από αυτές τις διατάξει. Δεν ισχύει αυτό, διότι ξέρουμε ότι οι πηγέ του ESM ε, είναι κάτι που εξασφαλίζουν τα κράτη-μέλη. Οπότε, από αυτή την έννοια, είναι λογικό η εθνική διακυβέρνηση να είναι καθοριστική σημασία στη διακυβέρνηση αυτού του οργανισμού, όπω ε, προβλέπεται από την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω, λοιπόν, ότι βάσει και του νέου προγράμματο του συνασπισμού τη γερμανική κυβέρνηση, θα ενσωματωθεί στο ενωσιακό δίκαιο η ΕΣΕΜ και ότι ενωμένοι θα στηρίξουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρί να χάσουμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα πρόοδου για να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε το πλαίσιο τη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκουαλτιέρη. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον επόμενο βασικό μιλητή για αυτήν την συνεδρία, τον κύριο Νόρμπερτ Μπράκμαν, μέλος Επιτροπής Προπολογισμού της Γερμανικής Bundestag. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι συνάδελφοι, ποιος είναι ο ρόλος ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων. Τρία σημεία θέλω να σχολιάσω. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε κάποιες προτάσεις στις 6 Δεκεμβρίου του 2017 και λέω ότι δεν ε, απαιτούνται αλλαγές ε, των συνθήκων. Αυτό ε, θεωρώ ότι είναι προβληματικό και από νομικής πλευράς, διότι υπερβαίνει η Κομισιόν κάποια όρια. Δεν μπορεί να παραγνωρίσει αυτά τα δισεκατομμύρια τα οποία προβλέπονται, 18 δις και έχουμε και 500 δις χωρίς να προτείνεται ε, δυνατότητα να εξουσιοδοτηθεί η ε, εκταμείευση αυτών των κονδυλίων και από τα κράτη. Έχουμε και το άρθρο 352 για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί αυτό το άρθρο να είναι η νομική βάση από νομική πλευρά, λοιπόν, οι προτάσει Κομισιόν δεν στέκουν, αλλά υπάρχουν και πολιτικά ζητήματα πολύ σοβαρά. Θα έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Νομισματική Ένωση. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντική πρόκληση η προσαρμογή ε, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, αλλά ε, όταν έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, δεν θα έχουμε και μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων δεν ε, πρέπει να έχουν λόγο και τα κράτη που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Θα πρέπει η συμπερίληψη του ταμείου, του ταμείου αυτού στην Ένωση να συνοδευτεί από αλλαγή της συνθήκης, κατά την άποψή μας. Και θα πρέπει να απασχολήσει τους πάντες αυτό το ζήτημα ότι μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θεσμικό όργανο, με πολύ μεγάλο όγκο, με σχηδαίες αρμοδιότητες και ευθύνες και λειτουργίες. Θα αναλάβει και τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξυγένσης. Θα πρέπει να είναι νομιμοποιημένο αυτό το νέο όργανο. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα επιβαρύνει ε, και θα συζητηθεί πολύ και στην προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογές. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα δεχθούν αυτές τις προτάσεις. Ε. Βέβαια μπορώ να μιλήσω μόνο για τη Γερμανική Βουλή. Εμείς ε, δεν θα φυστούμε προσπαθειών να έχουμε μια ενεργό συμμετοχή. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την ελπίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι τα κράτη-μέλη θα εκχωρήσουν ελαφρά την καρδία αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί ε, να υπάρχει ακριβώς υποχρέωση δημοκρατικής λογοδοσίας προς αυτά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν στέκει. Και σε ό,τι αφορά ε, την ε, χορήγηση των κονδυλίων, είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τους εθνικούς υπερπολογισμούς και τον ενωσιακό. Η Γερμανία τον Οκτώβριο του 2017 δήλωσε ότι είναι ε, το τελευταίο, η τελευταία ασφαλιστική δικλίδα αυτός ο ευρωπαϊκός ε, ε, μηχανισμό σταθερότητας και αποτελεί την έσχατη λίστα. Πρέπει να υπάρχει σίγουρα μία ευθύνη, αλλά αυτή θα πρέπει να παραμείνει ε, στα κράτη-μέλη εν τέλει. Τα κράτη-μέλη δηλαδή και τα εθνικά κοινοβούλια είναι αυτά τα οποία και στη συνέχεια θα πρέπει να έχουν τον τελευταίο λόγο και τον έλεγχο για την εκταμείωση των κονδυλίων αυτού του ταμείου. υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα στην ε, Γερμανία ότι συνδέεται με την ε, συμμετοχή του Γερμανικού Κοινοβουλίου η εκπροσώπησή μας ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, που σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αποφαίνεται ε, και αυτό τον κανόνα τον έχει κατοχυρώσει και το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο σε απόφασή του. Επομένως, συνταγματικό είναι ε, να μην ε, παραγνωρίζεται το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά ε, την νομιμοποίηση αυτού του νέου μηχανισμού. Και γι' αυτό η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την παροχή χρηματοοικονομικής βοήθειας αυτή οι αποφάσεις σχετικές να μην λαμβάνονται μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι εξασφαλισμένη η συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Το τρίτο σημείο είναι ότι φυσικά και η Γερμανία επιθυμεί την ε, ε, συνέχιση των προσπαθειών. Δεν θα προσπαθήσουμε να εμποδίσουμε την ε, μετάβαση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Σίγουρα όμω θα πρέπει να υπάρχει έλεγχο τη ισονομική πειθαρχία των κρατών μελών. Και θα πρέπει να δούμε τα ταμείο το διεθνές ε, τι προτείνει σε ό,τι αφορά την επίβλεψη και εποπτεία των ε, προγραμμάτων προσαρμογής. Ε, μέχρι τώρα είχαμε την Τρόικα. Τώρα θα έχουμε ένα νέο μηχανισμό. Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο ως Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο και να μην υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να είναι ανεξάρτητο όπως είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή ε, η Τράπεζα Επενδύσεων. Μόνο έτσι θα μπορεί να εξασφαλίσει ε, την ε, δημοσιονομική εποπτεία και να μην επηρεάζεται. Βέβαια η απόφαση σίγουρα θα ληφθεί εν τέλει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά τουλάχιστον θα είναι σαφές πού ε, ξεκινάει η πολιτική ευθύνη και πού λήγουν απλά οι οικονομικές αναλύσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μπράκμαν. Ο ρόλος στην κυρία Αλμπουκέρκη από την Πορτογαλική Βουλή, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Πορτογαλικής Βουλής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής, θέλω να θυμόμαστε ότι η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2007 εξελίχθηκε και μετατράπη σε μια κρίση κρατικού χρέους και μετά σε κρίση οικονομική και κοινωνική που έπληξε σοβαρά πολλές χώρες της Ευρώπης, της Ευρωζώνης και όχι μόνο. Ήταν η πρώτη μεγάλη κρίση εδώ και πολλά χρόνια και η πρώτη από την ε, δημιουργία του κοινού νομίσματος. Εκτέθηκαν αδυναμίες που υπήρχαν ήδη από την εποχή δημιουργίας του ευρώ. Ε, με την τεράστια πίεση της κρίσης και της μετέπειτα εξελίξης φτάσαμε σε μια Ευρώπη που πέρα από κάποια βραδύτητα παρόλα αυτά κατάφερε να δώσει αποκρίσεις για να ξεπεραστεί η κρίση και δημιούργησε θεσμούς και μηχανισμούς για να αντιμετωπιστούν κάποιες από τις ε, αδυναμίες που υπήρχαν από τον καταβολών του συστήματος. Έτσι φάνηκε ότι τα τελευταία χρόνια μπορούμε να κάνουμε πολλά παρά τις προφανείς δυσκολίες που φάνηκαν και από τις πρώτες παρεμβάσεις σε αυτό το πάνελ για να συμβάσουμε διαφορετικές ε, πολιτικές απόψεις, ε, διαφορετικές προοπτικές και ε, συγκεκριμένα προβλήματα που προκύπτουν από την τεράστια ποικιλομορφία που εκπροσωπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφέ ότι θα είχαμε συχνά καλύτερα αποτελέσματα αν μπορούσαμε να δράσουμε ταχύτερα. Όμω, επίση είναι αλήθεια ότι έγιναν πολλά. Και πολλά που απομένουν να γίνουν όμω. Γι' αυτό οφείλουμε να βελτιώσουμε τα όσα έχουν εξευρεθεί ω τώρα ω λύσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει προτάσει σε πολλού διαφορετικού τομεί και οι Ευρωπαίοι κρατών και κυβερνήσεων έχουν θέσει φιλόδοξου στόχου ε, και ε, ραντεβού στον χρονικό ορίζοντα για να δούμε ή όχι αν θα επιτευχθούν. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον βασίζεται πολύ σε κανόνε. Και χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο οργανισμού και φορεί, ακόμη και για λόγου ε, δημοκρατικού ελέγχου, λογοδοσία, accountability όπω λέγεται, ενώπιον όλων των πολιτών. Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η μετατροπή του Ευρωπαϊκού Μοχανισμού Σταθερότητα σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, ασχέτω του τίτλου που θα επιλεγεί. Ε, θα πρέπει να κοιτάξουμε αν μπορούμε να μετατρέψουμε ένα μηχανισμό στήριξη σε περιπτώσει κρίση σε ένα θεσμικό όργανο με περισσότερε αρμοδιότητε που θεσμικό να είναι πιο εύρωστο και δημοκρατικό ε, ε, ελέγξιμο, δυνατόν να ελεγχθεί από του εκπροσώπου των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι σημαντικό λοιπόν μεταξύ των νέων αρμοδιοτήτων που θα προβλεφθούν για αυτό το θεσμικό όργανο ένα ρόλο backstop στο Ταμείο Διάσωση ε, που μπορεί να υπάρχει. Αυτό είναι σημαντικό για να προχωρήσει η Τραπεζική Ένωση, παρόλο που δεν είναι το μόνο που λείπει από αυτήν. Να θυμίσω ότι το εγχείρημα τη Τραπεζική Ένωση πρέπει να ελέγξει το τι θα γίνει μεταξύ τη σύνδεση κεντρικών τραπεζών με τι υπόλοιπε και να μην υπάρξουν καταστροφικέ συνέπειε. Διότι μπορεί να υπάρξουν ε, πολύ επιζήμιε κοινωνικέ συνέπειε, εφόσον η σύνδεση αυτή δεν ελεγχθεί. Για τις συζητήσει στο ΕΚΟΦΗΝ τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την Τραπεζική Ένωση ήταν πάντα δυσχερή. και από την αρχή ακουγόταν η μέρημνα ότι πρέπει από τη μια να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνο και από την άλλη να διαιρεθεί ο κίνδυνο. Η μεταφορά τη κυριαρχία προ του προ τα θεσμικά όργανα που δημιουργείται. Ήταν ένα στοιχείο κινδύνου. Όμω ένα άλλο στοιχείο κινδύνου είναι ότι λείπουν ακόμη πολλά. Χρειάζεται λοιπόν να ληφθούν αποφάσει σε κεντρικό επίπεδο, αλλά να δούμε πώ οι, κίνδυνοι, οι αποφάσει αυτέ μάλλον μπορούν να αναλυθούν ω ευθύνε από του ε, φορολογούμενου των κρατών μελών. Η δημιουργία ενό Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου με ευθύνη backstop είναι ένα σημαντικό βήμα για να συμπληρώσουμε τον δρόμο που μας απομένει προς την βελτίωση αλλά θα πρέπει να έχουμε και σταθερούς στόχους με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να μπορούμε να προβλέψουμε στοιχεία όπως η εγγύηση των καταθέσεων. Το 2012, το 2013 είδαμε να επιτυγχάνουμε πολλά σχετικά, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε μια νέα κρίση, ώστε υπό το βάρο μια τέτοια κρίση να αναγκαστούμε να προχωρήσουμε ε, και να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση. Σε ό,τι αφορά την συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων, Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρότασή της ε, κάνει μια εύστοχη ένδειξη ε, με ενεργότερο ακόμη ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου που μας εκπροσωπεί όλους αλλά θυμίζω ότι πολλά από αυτά που αναλογούν ε, στην παρακολούθηση των εξελίξεων από τους πολίτες και τη συμμετοχή των πολιτών έχουν να κάνουν με τους κυβερνώντες της κάθε χώρας. Εκείνοι είναι υπεύθυνοι για τις αποφάσεις, για τις για την ε, διενέργεια των συζητήσεων και ενώπιον των κοινοβουλίων του, ενώπιον των πολιτών τη χώρα του, είναι υπεύθυνοι για την άμυνα των θέσεών του και για την προάσπιση αυτών των θέσεων. Γι' αυτό θα πρέπει αυτό ο θεμελιώδη ρόλο να αναγνωριστεί στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μην ξεχνάμε ότι σε πολλές χώρες οι κυβερνώντες ε, τείνουν να εξηλαιώνονται ενώπιον των πολιτών τους ε, ευθύνε ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο κεντρικό επίπεδο. Πρέπει να το προσέξουμε και αυτό. Η προθυμία των Ευρωπαίων ευθυνόντων να αποδώσουν κάποιες αρμοδιότητες και στα Εθνικά Κοινοβούλια είναι σημαντικό στοιχείο για να υπάρξει μεγαλύτερη εγκύτητα και σύγκληση. Όμως πρέπει ε, να δούμε τη σχέση ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και εθνικών κοινοβουλίων. Όλοι οι κυβερνώντε και στι χώρε μα είναι δημοκρατικά εκλεγμένοι, άρα έχουν τι δικέ τους ευθύνε εναντίον των δικών του κοινοβουλίων. Θα πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν σε αυτό το δρόμο, σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε και εμπόδια, όμω δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κρίση που στην πιο δύσκολη φάση τη έχει ξεπεραστεί, δεν σημαίνει ότι έχουμε ξεφύγει τελείως και ότι τα πάντα έχουν επιληθεί για να μην χειροτερέψουν τα πράγματα, θα πρέπει να βρούμε απαντήσει για όλε αυτέ τι ανησυχίε και να σκεφτούμε ότι αυτό που βοηθά του πιο αδύναμου μεταξύ ημών είναι συνολικά βοήθεια για την Ευρώπη, στο σύνολό τη. Ευχαριστώ. Благодаря ви, госпожо Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Αλμπουκέρκε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Λιμπεράτσκι για να συνεχίσει την, να προεδρεύει στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι έχετε αυτό το ροζ χαρτάκι. Να, πρέπει να το συμπληρώσετε αν μπορείτε για να απαντήσετε στην έρευνα. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή αυτή και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι θέμα της συνεδρίασής μας είναι η μετάβαση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας προς το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος των ε, κοινοβουλίων. Και ε, σε σχέση και με τα λεγόμενα από τον Ρομπέρτο, θα έχουμε απαντήσεις. Την απάντηση του κυρίου Μπάκμαν και την απάντηση της κυρίας Αλμπουκέρκε. Μόλις τώρα τις ακούσαμε. Έχω την εντύπωση ότι δεν τίθεται πλέον το ερώτημα το επαρξιακό εάν θα το κάνουμε, τίθεται το ερώτημα του τρόπου, πώς θα το κάνουμε για να έχουμε επιτυχία. Με όλα αυτά λοιπόν που ακούσαμε, με την έρευνα, με το ερωτηματολόγιο, έχουμε ε, κάνει μία ε, καλή προπαρασκευαστική δουλειά. Να δώσω το λόγο στην Αντιπρόεδρο Φαμπιέν Κέλλερ από τη Γαλλική Γερουσία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Λιμπεράτσκι που μου δίνετε το λόγο. Καταρχάς δύο σκέψεις θα ήθελα να εκφράσω διότι είμαι γερουσιαστής και μέλος της Επιτροπής Οικονομικών της Γαλλικής Γερουσίας. Πρώτον, θα ήθελα να αναφερθώ στη ζώνη του ευρώ και στην ανάγκη εμβάθυνσης του συντονισμού των πολιτικών, των οικονομικών πολιτικών στη ζώνη του ευρώ, σεβόμενοι πάντοτε πλήρως, αγαπητή κυρία Πρόεδρε στο τις χώρες που δεν έχουν ακόμα προσχωρήσει στη ζώνη του ευρώ. Θα ήθελα να θέσω το εξή ερώτημα. Δεν θα ήταν προτιμότερο να στηρίξουμε απερίφραστα ε, τη δημιουργία ενός προπολογισμού για τη ζώνη του ευρώ, ενός αυτόνομου προϋπολογισμού πέρα από την πρόταση της δημιουργίας μιας απλής δημοσιονομικής γραμμής, γραμμής στον προϋπολογισμό. Δεύτερο ερώτημα, η δεύτερη σκέψη που θα ήθελα να εκφράσω έχει να κάνει με το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Είναι μεγάλη χαρά για εμάς που είμαστε εδώ και συναντούμε τους συναδέλφους από τις άλλες χώρες. Είναι η τρίτη φορά που προσωπικώς ε, εγώ συμμετέχω σε μια τέτοια συνάντηση, αλλά θα πρέπει να συναντιόμαστε ακόμα πιο συχνά. Ο συντονισμός είναι απαραίτητος μεταξύ των εθνικών οικονομικών πολιτικών και ε, της πολιτικής που ασκείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχει και το θέμα της υπεράσπισης, της εξήγησης της ευρωπαϊκής πολιτικής στο ευρύ κοινό. Και η κυρία Αλμπορκέκε μόλις τώρα το ανέφερε. Θα πρέπει όλοι να, είμαστε, ε, να μεταλαμπαδεύουμε το μήνυμα των ευρωπαϊκών στρατηγικών, τις οποίες άλλωστε προσυπογράφουμε αφού βρισκόμαστε εδώ. Μιλούμε για τη δημιουργία ενός κοινοβουλίου της ζώνης του ευρώ. Όχι νέο όργανο, αλλά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, Έχω υπάρξει δήμαρχος στο Στρασβούργο και ελπίζω να με συγχαρήσετε, αλλά θα ήθελα να συνηγορήσω υπέρ της διοργάνωσης τέτοιου είδου συνεδριάσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα ε, στην πόλη του Στρασβούργου. Σας ευχαριστώ θερμά. Thank you very much. Madame, for such a very clear Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Κέλλερ, για την ε, πολύ σαφή σα δήλωση. Είναι ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης. Επόμενος ομιλητής είναι η κυρία Μαργαρίτα Μάρο από την Πορτογαλική Εθνοσυνέλευση. Αντιπρόεδρος της ε, Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η προαλή σας έθεσε ένα ερώτημα που δεν μπορούμε να καλύψουμε σε δύο λεπτά για ένα κοινοβούλιο της Ευρωζώνης, όμως θέλω να κάνω δύο ξεκάθαρες παρατηρήσεις. Πρώτον, ανάγκη μεγαλύτερου συντονισμού στην Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει ότι μια και μιλάμε για οικονομική διακυβέρνηση, η οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να ε, νοείται ως δημοκρατική διακυβέρνηση με δημοκρατικό έλεγχο. Αυτό είναι το σημείο αφετηρίας για να υπάρξει ένας περαιτέρω στοχασμός για τη μετατροπή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας σε Ευρωπαϊκό ε, Νομισματικό Ταμείο. Δηλαδή, αυτές οι αρχές του δημοκρατικού συντονισμού και του δημοκρατικού ελέγχου θα πρέπει ρητός να ε, εκφραστούν σε αυτή την προσπάθεια μετατροπής. Είναι σημαντικό ο μηχανισμός σταθερότητας να μετατραπεί σε Ευρωπαϊκό ταμείο, αλλά με μία ε, προοπτική ε, των όσων προβλέπουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Εδώ θα ήθελα να υποστηρίξω την ε, προοπτική που μας παρουσίασε περισσότερο ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ, ο κύριος Γκουαλτιέρη, από ε, αυτό που μας είπε ο κύριος Μπράκμαν. Δηλαδή, σε αυτή την προσπάθεια μετατροπής πρέπει να κοιτάξουμε να δημιουργηθεί ένας ευρωστότερος, πιο δομημένος και πιο ευέλικτος μηχανισμός, αλλά στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου. Όχι μια νέα διακυβερνητική συνθήκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη χαρά δίνω το λόγο στον κύριο Δημήτριο Παπαδημούλη, Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η πρόταση της Κομισιόν για τη μετατροπή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο είναι ένα βήμα προς τη θετική κατεύθυνση. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που έκανε ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Γκουαλτιέρη, ότι χρειάζεται να ενισχύσουμε και τη δημοκρατική λογοδοσία και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον έλεγχο αυτών των πράξεων. Δεν συμφωνώ με τις ε, ενστάσεις και τις διαφωνίες που κατέθεσε ο κύριος Μπράκμαν, γιατί πιστεύω ότι η εμπειρία μας διδάσκει ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπρος, κύριε Μπράκμαν. Όταν ξέσπασε η κρίση, που σημείωσε και η Πορτογαλίδα συνάδελφος, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε τους μηχανισμούς για να αντιδράσει. Και έφτιαξε καινούριου μηχανισμούς, όπως είναι ο ESM και πριν από αυτόν ο EFSF. Τώρα που τα πράγματα είναι πιο ήρεμα, πρέπει να προετοιμαστούμε για την επόμενη κρίση και πρέπει να ενισχύσουμε και την κοινοτική μέθοδο διότι η διακυβερνητική μέθοδος μόνη της έχει αποδείξει ότι είναι υπερβολικά δυσκίνητη και γραφειοκρατική και δεν μας προστατεύει από τη θύελα μιας μελλοντικής κρίσης. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερη ένωση στην πράξη και όχι στα λόγια. Φυσικά θα παίζουν ρόλο και τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά πρέπει να ενισχύσουμε και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγεται από τους πολίτες μας και πρέπει να κάνουμε βήματα και στην ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και στην ολοκλήρωση της Οικονομικής Ένωσης και στην ολοκλήρωση της Νομισματικής Ένωσης. Γιατί δεν είναι καλό για την Ευρώπη ο τρίτος πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι το Πανευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύσης Καταθέσεων που έχει προταθεί εδώ και δύο-τρία χρόνια από την Κομισιόν να μπλοκάρεται από λίγες κυβερνήσεις μέσα στο Συμβούλιο όπως είναι η Γερμανική και η Ολλανδική δεν μπορούμε να έχουμε μια Ευρώπη να τρέχει σαλαγός γρήγορα εκεί μόνο που συμφέρει τους ισχυρούς, τις πλούσιες χώρες, τις μεγάλες πολυεθνικές και να πηγαίνει πολύ αργά σαν το σαλιγκάρι ή προς τα πίσω σαν τον κάβουρα, σαν το καβούρι όταν μιλάμε για την κοινωνική πολιτική συνοχή, για την ολοκλήρωση τη Τραπεζική Ένωση, για την ενίσχυση τη δημοκρατική λογοδοσία. Και θέλω να πιστεύω ότι τέτοιε συναντήσει βοηθούν να κερδίζουν έδαφος απόψεις για περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Κράιταν Μπαρτόλο από τη Μάλτα, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θέλω να πω ότι το γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτό το ταμείο, ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο ίδρυση ενό τέτοιου ταμείου είναι ένα βήμα προ τα εμπρό. Και νομίζω ότι πρέπει να το επικροτήσουμε. Διότι είδαμε εκ των υστέρων ότι θα μπορούσαμε να είχαμε διαχειριστεί καλύτερα την ε, χρηματοπιστωτική κρίση αν υπήρχε ένα τέτοιο ταμείο όταν χτύπησε η κρίση. Και πιστεύω ότι ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι προετοιμασμένη σε περίπτωση που έχουμε μια νέα αντίστοιχη κρίση στο μέλλον. Δύο μικρές παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά καταρχάς ε, το όνομα του Ταμείου. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να το αποκαλέσουμε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Διότι η άποψή μου είναι πως αυτό είναι κάπως παραπλανητικό, καθότι έχει διαφορετικές, θα έχει διαφορετικές λειτουργίες από αυτές ε, που αποδίδουμε ή που έχει τέλος πάντων το Διεθνές Νομισματικό Όνομα, θα πρέπει να έχει διαφορετικό όνομα. Και κάτι πιο σημαντικό, επειδή η που εχει τελος παντων το διεθνες νομισματικο αρα θα πρεπει να εχει διαφορετικο ονομα και κατι πιο σημαντικο επειδη η χωρα μου είναι από τις μικρότερες χώρες ε, τη. Ευρωζώνης, παρότι πηγαίνει πολύ καλά ε, από άλλες μεγάλες χώρες, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει η δικαιωματική δομή του ESM και να χρειάζεται ομοφωνία για όλες τις αποφάσεις. Να παραμείνει δηλαδή το ισχύον σύστημα της ομοφωνίας. Επίσης, ό,τι αφορά το ενδεχόμενο της χρήσης του νέου ταμείου. Ας το πούμε Ευρωπαϊκό Νόμισμα το προς το παρόν. Να είναι η τελευταία ε, ασφαλιστική δικλίδα, αλλά αυτό πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο για να κατανοήσουμε σε βάθος τις επιπτώσεις που θα είχε κάτι τέτοιο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ γιατί σεβαστήκατε όλοι και το χρόνο αγόρευσης. Επόμενος ο Πέτερ Όμτσικ, μέλος Επιτροπής ε, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων από την Ολλανδία. Επίσης, παρακαλώ για το σκάμερα για να μπορούν να σας εντοπίσουν, να σηκώνετε το χέρι σας πριν πάρετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ για τα πολύτιμα σχόλια. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω δύο-τρία σημεία για να υπερασπιστώ τον κύριο Μπράκμαν, τον οποίο ε, υποστηρίζω σε αυτά που είπε. Πρώτα απ' όλα, επειδή ακούσαμε τον κύριο Τομπρόφσκι το πρωί, που είπε ότι θα έχουμε μια πλήρη ονέ μόνο εάν είναι δημοκρατική αυτή η ονέ. Έχει δίκιο ο κύριο Τομπρόφσκι κατά την απόψη μου. Όμω 26 κοινοβούλια προσχώρησαν ε, στην πρωτοβουλία του Ολλανδικού Κοινοβουλίου για την υπογραφή μια δήλωση, μια επιστολή προ το Συμβούλιο Υπουργών και προ τον πρόεδρο του Eurogroup, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στα έγγραφα. Διότι προς το παρόν δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ε, ε, κατάρτιση νομοθεσίας και την λήψη αποφάσεων εντός του Eurogroup. Και ελπίζω να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε γι' αυτό από κοινού, γιατί οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνουμε θα πρέπει εμείς ως βουλευτές να μπορούμε να ελέγχουμε τις αποφάσεις αυτές, ιδίως όταν αφορούν σε εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, ανησυχώ, ανησυχώ γιατί υπάρχει ένα τεράστιο κίνδυνο τον οποίο έλαβε η ΕΚΤΑ. Χωρίς 2,5 2,5-4 εκατομμύρια ομόλογα. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Έξι χρόνια έχουμε ανάπτυξη, αλλά συνεχίζεται αυτή η πολιτική. Είναι μια επικίνδυνη πολιτική. Εάν τώρα θεωρούμε ότι μπορούμε την κρίση να την με τέτοια πήγοντα ε, κονδύλια τα οποία ε, ποιος θα τα αποπληρώσει και τα οποία θα δημιουργήσουν μια πιο άσχημη συστημική κρίση, είμαστε σε λάθος δρόμο. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να δημιουργήσουμε θεσμικού, θεσμούς που δεν θα αυξάνουν αλλά θα μειώνουν τους συστημικούς κινδύνους. Και αυτό ίσως με την κατάργηση αυτού του προγράμματος της ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤΑ. Να μην έχουμε αυτά τα τεράστια κονδύλια. Γιατί τα κράτη είναι αυτά που έχουν την πρωταρχική ευθύνη και πρέπει να λύσουν το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο κ. Μπέρντ Λούκε, με βάση τον κανόνα μας, δύο εθνικοί βουλευτέ, ένα ευρωβουλευτής. Ευρωβουλευτής από το Γερμανίο, κύριο Σελούκε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω γερμανικά. Πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά την παρέμβαση του κυρίου Γκουαλτέρη και του κυρίου Παπαδημούλη. Ε, θα ήθελα να διαφωνήσω διότι νομίζω ότι αυτό που λέγεται ε, κυρίως ε, είναι η σχέση μεταξύ ευθύνης και υπευθυνότητας λογοδοσίας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αν θέλουμε να έχουμε μια οικονομία που να λειτουργεί εύρωστα και εύρυθμα να μην τα μπερδεύουμε αυτά τα δύο. Ο κύριος Γκουαλτέρη... Ε, έκανε κάποιες ε, προτάσεις και ε, μας είπε ότι υπάρχουν κάποιες προτάσεις και από τον ακαδημαϊκό κόσμο. Ε, ότι δεν θα πρέπει σε ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση του χρέους ε, να ε, υπάρχει αυτός ο ρόλος για το ταμείο. Εγώ νομίζω όμως ότι αυτό ακριβώς χρειάζεται, δηλαδή θα πρέπει αυτό το ταμείο να εγκρίνει δαπάνες και βοήθεια μόνο όταν η κατάσταση της χώρας μπορεί να είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα σε ό,τι αφορά το χρέος. Αν το χρέος δηλαδή είναι βιώσιμο, ε, τότε ε, υπάρχει αυτό το πρόβλημα της ανάγκης δηλαδή αναδιάρθρωσης, ε, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να επιβαρύνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι αναλύσει αυτής της βιωσιμότητας του χρέους να μην ε, είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιρροών ε, στο βαθμό που είναι μέχρι τώρα. Ε, και σε αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, θα πρέπει να κάνει αυτές τις αναλύσεις βιωσιμότητας αλλά αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό που ε, κάνει η Κομισιόν. Δηλαδή η Κομισιόν είναι αυτή που έχει αναλάβει μέχρι τώρα την ανάλυση της βιωσιμότητας. Θα πρέπει λοιπόν να, να έχουμε αυτό το ανεξάρτητο θεσμικό όργανο που θα μπορεί να είναι αρμόδιο για τη βιωσιμότητα του χρέους και δεν θα πρέπει να υπόκειται ή να υποβάλει σε κανέναν πολιτικό ε, σε καμία πολιτική επιρροή αυτό το θεσμικό όργανο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, και τώρα ο κύριος Μανιός, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων από την Ελλάδα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Εκτιμώ, παρότι δεν είμαι οικονομολόγος, ότι η μετατροπή του ESM σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα είναι ένας σταθμός στην ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι ένας μοχλός μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών της. Ακούστηκε ότι μπορεί το Νομισματικό Ταμείο να συντελέσει στην δημιουργία της Ευρώπης των δύο ταχυτήτων. Δεν ξέρω πόσες ταχύτητες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν φταίει το ευρώ από μόνο του αν υπάρχουν δύο ή περισσότερες ταχύτητες. Οι πολιτικές που ακολουθούνται δημιουργούν το, το τεράστιο ηθικό και πολιτικό ζήτημα για την ύπαρξη ευρωζώνης ανάμεσα στις ανισότητες που υπάρχουν και μέσα στα μέλη και ανάμεσα στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι πολιτικές είναι η λύση του προβλήματος των ανισοτήτων. Ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο που θα είναι γέννημα του ευρωπαϊκού κεχτημένου που λέμε δεν θα έχει κανένα από τα χαρακτηριστικά και τις νοοτροπίες που είχε και έχει το δούνου του. Έχουμε το εξαιρετικά αρνητικό παράδειγμα της παρουσίας του δούνου του στην Ευρώπη. Θα μιλήσω μόνο για τη χώρα μου, για την Ελλάδα τι ήταν οι προτάσεις του Δούνου Ήταν έξω από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων, ε, εξευθελιστικές ε, περικοπές των δαπανών και στο τέλος τι μας είπαν ότι έκαναν λάθος με αυτή την πολιτική και δεν πέτυχε η συνταγή τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να πάρει αυτή την ιστορική ευθύνη που της αναλογεί. Να δημιουργήσει αυτό το εργαλείο που θα μπορεί να προβλέπει και να διορθώνει τα λάθη που συμβαίνουν και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα η κυρία Μπίρκετ Παρσάκ από την Bundestag και την Επιτροπή Προπολογισμών. Jetzt. Okay. Αξιότιμε Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, σε ό,τι αφορά την ομάδα FD, σε ό,τι αφορά την μετατροπή του Ταμείου Σταθερότητας, μάλλον του Μηχανισμού Σταθερότητας ε, σε ένα ε, νομισματικό ταμείο. Εμείς θεωρούμε ότι με βάση την ομολογία του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου την απόφαση της Λισαβόνας όπως λέγεται πρέπει να κυριαρχεί η αρχή της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου ό,τι αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο του προπολογισμού. Δεν μπορεί να αντικαταστηθεί ο Εθνικός Κοινοβουλευτικός Έλεγχος από ε, τον έλεγχο που θα γίνεται μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι μιλάμε για ε, ένα ζήτημα καθορισμού της ταυτότητας και ε, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό για το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο. Δεν μπορεί να είναι αρμοδιότητα, παραδείγματο χάρη, μόνο ε, τη Ευρώπη, χωρί να έχει λόγο ο γερμανικό λαό μέσω του κοινοβουλίου του. Και σε ό,τι αφορά αυτά που είπε ο κύριο Μπράκμαν, έχουμε το άρθρο 352 που θεωρείται νομική βάση από το δικαστήριο. Το 98 ήδη ε, θεωρήθηκε αυτό το άρθρο ότι ε, είναι περιοριστικό ε, σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περιορίζεται δηλαδή ε, η αρμοδιότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και επίσης υπάρχουν οικονομολόγοι οι οποίοι έχουν μιλήσει και εκφραστεί. Είχαμε ε, και από τη Γερμανία εκφράσει τις επιφυλάξεις μας απέναντι στην ΕΚΤ σε ό,τι αφορά ε, τα ποσά αυτά ε, τα οποία δίνονται και τα οποία πραγματικά υπερβαίνουν σχεδόν τον όλο γερμανικό προϋπολογισμό. Είναι σημαντικά ποσά και δεν μπορώ βέβαια να αναλύσω ακόμη περισσότερο ε, τις οικονομικές και νομικές διαστάσεις και παραμέτρους, αλλά ε, σίγουρα δεν πρέπει να ε, πριονίσουμε την καρέκλα πάνω στην οποία καθόμαστε. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει γερμανική νομολογία, αλλά υπάρχει και η ευρωπαϊκή νομολογία, την οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη γιατί από αυτές τις αποφάσεις φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί των ευρωπαϊκών αρμοδιοτήτων. Δεν πρέπει να καταργηθεί αυτή, αυτός ο περιορισμός. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαλεώτη από την Ιταλική Γερουσία. Thanks, Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω το πώς θα ονομαστεί το νέο θεσμικό όργανο, αυτό που θα προκύψει από τη μετατροπή του ESM, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα, είναι θεμελιώδου σημασία. Διότι σε σχέση με όσα μα είπε και ο κύριος Γκουαλτιέρη και όσα μα έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο δεν είναι καταλληλό, ο καταλληλότερο τίτλο. Αν ακούσουμε και το γερμανό συνάδελφο Μπράκμαν, νομίζω ε, ότι μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο ταμείο. Όμως η δική σας πρόταση είναι αντιδιαμετρικά αντίθετη από αυτήν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διότι είναι σαφές, από όσα λέτε, ότι θέλετε να μεταφερθούν οι ευθύνε για τη διαχείριση κρίσεων και τη διαδεδότηση στο νέο ταμείο. De facto λοιπόν θα ανακληθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο να εντοπίζει τις ε, ε, ελλείψεις ισορροπίας μακροοικονομικός και να ε, ορίζει προγράμματα ενίσχυσης και το πώς θα υλοποιηθούν. Άρα φαίνεται να γίνεται σαφές ότι η διενειοδότηση από το νομισματικό ταμείο θα πρέπει να γίνει κανόνας για τις χώρες που κινδυνεύουν να μην έχουν πρόσβαση στις αγορές με όλες τις παράπλευρες συνέπειες το, της αναδιάρθρωσης. Μιλάμε για μια πολύ διαφορετική πρόταση σε σχέση με τη νέα λειτουργία του νέου μηχανισμού σταθερότητας και για την κυβέρνηση. Ε, στο κάτω-κάτω της γραφής δεν είναι τόσο πολύ το θέμα του ελέγχου των Εθνικών Κοινοβουλίων μόνο είναι ότι το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο με τη γερμανική πρόταση, τέλο πάντων αυτά που εσείς είπατε, θα είναι υποχείριο των χωρών πίστοσης. Δηλαδή, από αυτήν την οπτική γωνία είναι τελείως ασαφές πως αυτό θα φέρει περισσότερο δημοκρατικό, περισσότερο δημοκρατικό έλεγχο και λογοδοσία ε, προς το, από το Ευρωκοινοβούλιο και από τα εθνικά. Θα ήθελα λοιπόν να μας το εξηγήσετε λίγο παραπάνω, διότι να, να δούμε αν καταλάβαμε ε, τη θέση σας. Και αυτό σε αντιπαραβολή με την άλλη θέση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ο κατάλογος των αγοριτών εκ μέρους των Εθνικών Κοινοβουλίων εξυνλήθη. Θα παρακαλέσω λοιπόν όλους αγορητέ που τοποθετήθηκαν εν είδη εισαγωγή να σχολιάσουν όσα ακούστηκαν ή να μα πούν ότι θεωρούν ότι είναι απαραίτητο σε αυτή τη φάση. Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ χρήσιμη και οικοδομητική συζήτηση και δείχνει την ε, προτεθέμενη αξία αυτής της διακοινοβουλευτικής ε, συνόδου που φέρνει στον ίδιο χώρο εθνικούς βουλευτές και και ακούμε τις δικές τους προοπτικές, τη δική τους ερμηνεία με μια προσπάθεια να υπάρξει μια μηδέα κατανόηση. Να σχολιάσω ιδίω για αυτά που είπε ο κύριος Μπράκμαν. Διότι όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, Είμαστε μάλλον σε, μια σε ένα διαφορετικό μήκο κύματο. Κατά τη δική μου την άποψη υπάρχουν κάποιε παρερμηνίε ή ίσω εγώ να μην κατέλα, κατάλαβα καλά, να υπάρχει κάποια παρανόηση. Όπω είπε ο κύριο Μπράκμαν. Ε, βεβαίω υπάρχει ένα θέμα καθηκόντων, αρμοδιοτήτων, το τι θα αποδοθεί σε αυτό το θεσμικό όργανο. Και εδώ βλέπω να υπάρχει διαφωνία. Διότι βεβαίω αυτό που προτείνει ο κύριο Μπράκμαν να ανατεθεί στο νομισματικό ταμείο ένα ρόλο, ένας ρόλος που τώρα τον έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι που της αναθέτει η ίδια η συνθήκη η μακροοικονομική εποπτεία, η δημοσιονομική εποπτεία, ο σεβασμός των διατάξεων της συνθήκης και η παρακολουθήση, το να αποδοθεί κάτι τέτοιο στο νομισματικό ταμείο θα ήταν κάτι τελείως διαφορετικό και πολιτικό δεν ξέρω αν θα ήταν επιθυμητό, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπόλογη, ελέγχεται από το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο. Ένα ανεξάρτητο σώμα τώρα που σχεδιάζει τις οικονομικές πολιτικές και ε, έχει τόσο βαθιές ευθύνες που επιβάλλει τον σεβασμό της δημοσιονομικής πειθαρχία είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την οικονομική διακυβέρνηση και αυτό μάλιστα θα πετούσε ε, ευρύτερε αλλαγέ. Πρέπει να αλλάξουν τα άρθρα τη συνθήκη που αναθέτουν αυτή την ε, αρμοδιότητα, αυτό το καθήκον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και να πάρουμε αυτή την ευθύνη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να την πάμε σε ένα άλλο σώμα, σημαίνει ότι γίνεται μια ριζοσπαστική αναθεώρηση των συνθήκων μα. Πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκε, να γίνουν δημοψηφίσματα στα κράτη-μέλη. Ειλικρινώ λοιπόν μιλάμε για κάτι το άπιαστο. Άρα, ή δεν αλλάζουμε τίποτα και αφήνουμε τον ε, μηχανισμό σταθερότητα ω έχει, κάνουμε μια μικρή διακυβερνητική συνθήκη για να προσθεθεί το backstop. Διότι ειλικρινώ δεν καταλαβαίνω, ε, δεν νομίζω ότι κανεί σε αυτή την αίθουσα θεωρεί ρεαλιστικό να ε, συλλάβουμε ούτε καν ω προπτική μια τέτοια ριζοσπαστική αναθεώρηση των συνθήκων. Θα ήταν σφάλμα. Θα πάρουμε τώρα τι μακροοικονομικέ αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα τι αναθέσουμε σε αυτό το σώμα, αλλά πέραν από αυτό. Είναι τόσο μη ρεαλιστικό να, να έχουμε μια βαθιά αλλαγή, τόσο βαθιά αλλαγή στι συνθήκε. Δεν είναι καν σημείο που συζήτηση. Δεν είναι επιτάπητο. Τι είναι λοιπόν αυτό που έχουμε μπροστά μα, ε, επιτάπητο. Είναι αν θέλουμε να ε, πάρουμε κάποιες αρμοδιότητες και να τις προσθέσουμε στον ESM. Το backstop, την δυνατότητα να ε, δράσει ε, από μόνο του το Ταμείο, χωρίς τη συνδρομή του διεθνού Νομισματικού Ταμείου, να ζητήσει αναδιάρθρωση, διότι αυτή τη στιγμή ο μηχανισμός σταθερότητα την έχει αυτή τη ε, δυνατότητα. Αυτό που συζητάμε στην ουσία και λέμε όλοι είναι το να περάσουμε από το ε, κάτι που ενδυνάμει μπορεί να γίνει σε μια υποχρέωση. Δηλαδή όλες οι κεντρικές τράπεζες, όσοι ασχολούνται με το κρατικό χρέος, ξέρουν ότι εάν κάποιο μετατρέψει μια δυνατότητα σε υποχρέωση, είναι κάτι το θετικό και χαρνητικό. Με... Που προσθέτει κάποιο μια υποχρέωση σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη πίεση στην αγορά και ε, μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερο spread. Άρα ε, μπορεί να παραμείνει μια επιλογή, να μην είναι υποχρέωση. Είναι λογικό αυτό. Αλλά πέραν αυτού, γιατί θα είναι πιο αποτελεσματικό να γίνει αυτό μέσω του άρθρου 352 και όχι με τη διακυβερνητική μέθοδο. Πρώτον, θέλω να το πω αυτό στον κύριο Μπράκμαν, Λέτε ότι πρέπει να συμμετάσχουν τα κράτη-μέλη στη διαδικασία λήψη αποφάσεων, ακόμη και τα κράτη εκτό Ευρωζώνη. Μα αυτό λέει η διαδικασία 352. Ομοφωνία και από τα 28 κράτη-μέλη. Ακριβώ αυτό το πρόβλημα που ε, θέτεται, επιλύεται με τη διαδικασία του άρθρου 352. Και ορθώ είπατε ότι τα εθνικά κοινοβούλια εφόσον ε, ε, μπορούν να ελέγξουν δημοκρατικά τις κυβερνήσεις τους, ε, έχουν ένα τέτοιο ρόλο. Αυτό κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό που, κάνει, που γίνεται τώρα στη Γερμανία. Η κυβέρνηση ως προ τον ESM είναι υπόλογη ε, στην Bundestag, στην Ομοσπονδιακή Βουλή. Αυτό θα ισχύει. Δεν αλλάζει γιατί μπαίνει στη μέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλώ προσθέτει πάνω από την υπάρχουσα λογοδοσία, τον Δημοκρατικό Έλεγχο των Εθνικών Κοινοβουλίων, που δεν αλλάζει σε τίποτα, προσθέτει επιπλέον πλαίσιο λογοδοσία. Όχι απλώ δηλαδή δημοκρατικό έλεγχο από το Κοινοβούλιο προ τη δική του μόνο κυβέρνηση, αλλά τα εθνικά κοινοβούλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν τη δυνατότητα να ε, ζητήσουν ε, να ελέγξουν δημοκρατικά όχι μόνο το κράτο, το, την κυβέρνηση τη χώρα του, αλλά οποιονδήποτε στο, που συμμετέχει στον ESM. Δηλαδή μπορεί να τον καλέσουν στην Εθνική τους Βουλή και να συζητήσει και να δώσει αναφορά ω προ τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τίποτα δεν αφαιρεί από τι τωρινέ εξουσίε των Εθνικών Κοινοβουλίων. Προσθέτει κιόλα. Προσθέτει επιπλέον αρμοδιότητα, επιπλέον εξουσία να συμβάλλουν στο να διατηρηθεί η λογοδοσία για ολόκληρον τον ESM και όχι μόνο ω προ τον εκπρόσωπο του επιμέρου κράτου. Αυτό το βρίσκω θετικό. Θετικό είναι, διότι το ίδιο μπορεί να κάνει και το Ευρωκοινοβούλιο, α πούμε, και αυτό είναι θετικό. Μπορούμε να συζητήσουμε με τον κύριο Ρέγκλινγκ, μπορούμε να οργανώσουμε ακρόαση για τον ε, μηχανισμό σταθερότητα και να δούμε πώ θα πάει κτλ. Άρα, μιλώντα μεταξύ μα, νομίζω ότι κάποιε φορέ καταλαβαίνόμαστε, αλλά κάποιε φορέ υπάρχει περισσότερη παρανόηση παρά διαφωνία. Διότι, όπω έλεγα, το Ευρωκοινοβούλιο ενώ συμφωνεί με τη συμπερίληψη όλων αυτών στη συνθήκη, δεν έχει πουθενά αντίρρηση στην ειδική ευθύνη και εξουσία των Εθνικών Κοινοβουλίων και Κυβερνήσεων. Ε, Βεβαίω, δική του είναι η πόρη του ESM. Αλλά για τον ε, στόχο 2 και το ECBQE δεν ξέρω και την ποσοτική χαλάρωση δεν ξέρω ε, κατά πόσον αυτό είναι τώρα να το συζητήσουμε θέμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ε, ανεξάρτητη και βεβαίω η νομισματική πολιτική είναι κάτι το άσχετο, αλλά δεν έχει να κάνει με τι πολιτικέ αποφάσει. Ούτε με τον ESM και τη μετατροπή του σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Τέλος, είναι ε, αλήθεια ότι η αναγγελία περί ανανεωμένου μηχανισμού σταθερότητας, τα ε, οδηγήσει σε περισσότερη ολοκλήρωση και ένωση ε, μεταξύ των οποίων και τη δημοσιονομική δυνατότητα που έχουμε. Δηλαδή αυτό που είπαν οι συνάδελφοι, τον ευρωπαϊκό, τον ενωσιακό προπολογισμό. Ε, αλλά γιατί η νέα δυνατότητα που θα έχουμε δεν είναι κάτι που αυτομάτω προσφέρεται εφόσον εγκριθεί η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει την λειτουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα ω έχει αλλά προβλέπεται μια νέα δυνατότητα για το μέλλον και σε πολλές περιπτώσεις κάθε κάτος μέλος θα έχει δικαίωμα λόγου και άρνηση κυρίας. Ενώ λοιπόν ε, το να το κάνουμε αυτό δεν θα μας εμποδίσει από ένα βήμα πρόοδου, ενώ αν δεν το κάνουμε σίγουρα δεν θα έχουμε βήμα πρόοδου, αλλά και πάλι όσοι διαφωνούν με το βήμα πρόοδου δεν προσυπογράφουν αυτομάτως την, αλλαγή, στηρίζοντα την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλο πάντων, για να ολοκληρώσω, βρίσκω την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ε, μηχανισμό σταθερότητα ή νομισματικό ταμείο, όπω θέλετε να το πείτε, πολύ ισόρροπη. Και αν δούμε όλε αυτέ τι πτυχέ, καθώ και τη νομική βάση και τα εξετάσουμε προσεκτικά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι μια ε, συμβαστική πρόταση που πετυχαίνει το σωστό σημείο ισορροπία. Και ξεπλάγει κάπω, γιατί διάβασα το πρόγραμμα του γερμανικού συνασπισμού, που νομίζω είναι πολύ σαφέ και πηγαίνει σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα ακούω μια τελείω διαφορετική ερμηνεία από τον κύριο Μπράκμαν που ήταν και μέρο των συζητήσεων για τον συνασπισμό. Είναι θετικές οι δύο αυτές προτάσεις στη δήλωση, στο πρόγραμμα του συνασπισμού ε, των γερμανικών πολιτικών δυνάμεων. Εγώ έτσι τις είχα κατανοήσει. Ευχαριστώ πολύ τον ε, Πρόεδρο κύριο Γκουαλτιέρη για τα σχόλιά του και τώρα θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Νόρμπερτ Μπράκμαν να πάρει το λόγο. Να ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε μέσω τη συζήτηση, νομίζω ότι κατέστη προφανές ότι υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις ε, για τους στόχους που θα είχε ένα τέτοιο ταμείο νομισματικό, όπως αλλιώς το αποκαλέσει κανείς. Μετά την χρηματοπιστωτική κρίση, την κρίση χρέους, ε, υπάρχει με τον ε, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας αυτός ο μηχανισμός ανάληψης ευθύνης ε, και κάλυψης ουσιαστικά του χρέους. Πρέπει να δούμε όμως τι θα γίνει σε περίπτωση που επαναληφθεί η κρίση. Τι πρέπει να κάνουμε και αυτό το ρόλο τον έχει προς το παρόν το ESM. Τώρα όμως συζητάμε για τον στόχο και το πηγαίνουμε σε κάτι διαφορετικό που δεν είναι η ε, κάλυψη αυτή, αυτού του κινδύνου, αλλά μιλάμε για μακροοικονομικά προγράμματα αποτροπής κρίσεων, μιλάμε για την ε, εξομάλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και διαφορών στην Ευρώπη. Και εκεί μιλάμε για τη δυνατότητα δανεισμού, η βοήθεια που αυτό θα πρέπει να γίνεται σε εθνικό επίπεδο και το ε, θέτουμε υπό αμφισβήτηση. Επομένως το θέμα είναι η στοχοθέτηση. Ποιοι είναι οι στόχοι της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πούμε ότι, ε, όπως είπε και η κυρία Κέλλερ από τη Γαλλία, αν κάποιος θέλει ε, ένα νέο ε, καθήκον, ε, θα πρέπει να υπάρχει άλλη αλληλεγγύη για την κάλυψη, την οικονομική αυτού του καθήκοντος. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσω του πολιτισμού οικονομικού πλαισίου ή θα πρέπει να υπάρξει μια άλλη ενίσχυση του σχετικού προγράμματος. Δεν θα πρέπει όμως ε, να αντιμετωπίσουμε, να βάλουμε σε κίνδυνο αυτό το σύστημα, διότι υπάρχουν ε, σημαντικά ποσά τα οποία τίθεται σε κίνδυνο και έχουμε την εθνική ευθύνη των κρατών μελών. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε όλα αυτά στην αγορά γιατί θα προκαλέσουμε νέες κρίσεις ουσιαστικά. Αυτό το λένε οι Βρετανοί bad economics make bad policy, δηλαδή τελικά με τα μέσα τα οποία εμείς τα έχουμε ως ασφάλεια αν θέλετε θα δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα αντί να το λύσουμε. Κάποιος αναφέρθηκε στη συμφωνία του γερμανικού συνασπισμού. Πρέπει να τη διαβάσει κανείς ε, προσεκτικά. Γιατί συγκεκριμένα οι εταίροι ε, δεν συμφώνησαν πάνω σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό και η διατύπωση είναι συγκεκριμένη. Δεν λέω ότι στηρίζει η γερμανική κυβέρνηση. Γίνεται λόγος εκεί για το ενωσιακό δίκαιο, ε, την ε, τήρηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και αυτό συνιστά ένα σημαντικό περιορισμό. Και σίγουρα ε, στη Γερμανία τουλάχιστον πρέπει να γίνει τεράστια συζήτηση για το όλο αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ Κύριε Μπράκμαν, επόμενος ομιλητής η κυρία Μαρία Λουίς Αλμπουρκέκε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με ορισμένους από τους προλαλήσαντες, κυρίως με τον κύριο Κουαλτιέρη. Και πιστεύω ότι και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ισορροπημένη και καταλαβαίνω ότι πράγματι είναι δυνατό να προσπαθήσουμε να βάλουμε πράγματα που ακόμα δεν υπάρχουν. Όμως, σε κάποια σημεία έχουμε μείνει στο 12 και στο 13 δεν έχουμε προχωρήσει. Οι ίδιες ανησυχίες είναι παρούσες, οι ίδιες υποψίες ακόμα υπάρχουν για το τι θέλει να κάνει η Κομισιόν με την πρόταση αυτή. Οι ανησυχίες που εκφράζονται δεν είναι διαφορετικές από αυτές που εκφράζονταν το 2012. Η εμπλοκή, η συμμετοχή του Δούνου του ήταν αναγκαιότητα γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Δεν ήμασταν έτοιμοι να υιοθετήσουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να στηρίξουμε τις χώρες που αντιμετώπισαν δυσκολίες. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να ήμασταν σε θέση να τα κάνουμε από μόνοι μας αυτά. Δεν λέω να μην αναζητούμε τη στήριξη του Δουνουτού και εμείς είμαστε μέλη στο Δουνουτού ούτως ή άλλω, όλες οι χώρες νομίζω, και οι χώρες που αντιμετώπισαν προβλήματα, όμως είμαστε Ευρωπαίοι, είμαστε ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να προσπαθούμε να δρούμε εντός των συνθηκών μας, εντός των θεσμικών μας οργάνων, εντός των φορέων μας. Συμφωνώ με τον κύριο Γκουαλτιέρη, υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις εδώ και υπάρχουν και κάποιες προκαταλήψεις, κάποιες προηλημένες ιδέες και αντιλήψεις για τη σχέση μεταξύ πιστωτών και οφειλετών. Και αυτό οφείλεται, είναι αποτέλεσμα της κρίσης και των αρνητικών αντιδράσεων που έχουν υπάρξει στην κοινή γνώμη και στην πλευρά των πληρωτών και στην πιστωτών και στην πλευρά των οφειλετών. Υπάρχει αυτό το blame game, το παιχνίδι αλληλοκατηγοριών που εκτοξεύονται. Θα πρέπει να διαλύσουμε αυτές τις ανησυχίες. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι αν εμείνουμε σε αυτές τις προκαταλήψεις, σε αυτές τις προκαθορισμένες ιδέες που έχει ο ένας για τον άλλον. Δεν θα προχωρήσουμε αρκετά γρήγορα, δεν θα κάνουμε τα πάντα για να προλάβουμε μια επόμενη κρίση. Εάν, όπως είπε και ο κύριος Γκουαλτιέρη, πρέπει να επιταχύνουμε από τη δυνατότητα στην αναδιάρθρωση, στην υποχρέωση αναδιάρθρωσης, ξέρουμε πώς αυτά στις χρηματαγορές γίνονται ξαφνικά ε, αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Όταν το βάλουμε αυτό γραπτά και κάνουμε τις χώρες να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, τότε αυτό θα γίνει υποχρεωτικός, σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Όταν υπάρχουν θέματα βιωσιμότητας, πρέπει όλοι να καταλάβουν πόσο μεγάλη πρόοδο έχουμε σημειώσει, πόσο έχουμε προοδεύσει, πόσο πιο ασφαλείς είμαστε σίγουροι σήμερα ε, συγκριτικά με την κατάσταση πριν από κάποια χρόνια. Τώρα, προσπαθώντας να ενισχύσουμε, να θωρακίσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο και εάν σε αυτή την προσπάθεια συμβάλλουμε και βάλουμε στοιχεία που τελικά θα ε, επιταχύνουν την έλευση νέας κρίσης, θα γίνει αυτοεκπληρωμένη προετία, προφητεία και θα πρέπει να διαχειριστούμε μια νέα κρίση και πάλι. Μιλούμε για τις πολλαπλές ταχύτητες και τελικά θα υπάρχουν τόσες πολλές και διαφορετικές ταχύτητες που κάποιοι θα μείνουν οριστικά πίσω και αυτό θα είναι πολύ δυστυχές και θα είναι τελείως αντίθετο με αυτό που έχουμε προσπαθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, είτε υπάρχουν παρανοήσει, είτε υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές απόψεις και βεβαίως πάντοτε σέβονται όλοι όλες τις πολιτικές απόψεις. Ανεξαρτήτως τη αιτία, το σημαντικό είναι να έχουμε μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση. Δηλαδή, στην πρόταση της Επιτροπής να μην κυνηγάει κανείς ανεμόμυλος, να μην λέει ότι βλέπει πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα μέσα στην πρόταση και αν χρειάζεται η Κομισιό να το γράψει πιο ξεκάθαρα, ε, τότε ας το γράψει πιο ξεκάθαρα για να μην υπάρχουν συνέχεια αυτοί οι αβάσιμοι φόβοι και αβάσιμες ανησυχίες. Είναι οι ανησυχίε που κυρίω ανέφερε εδώ ο κύριο Μπράκμαν. Αλλά αν αυτό πιστεύει η Γερμανική Βουλή, η μέρο τη Bundestag τη Γερμανική Βουλή, ε, να το λύσουμε αυτό. Να διαλύσουμε αυτέ τι αβάσιμε ανησυχίε, να το διατυπώσουμε πιο ε, σαφώ. Και το θέμα τη δημοκρατική λογοδοσία, που είναι και το βασικό μα, να, να το πούμε ξεκάθαρα. Η λογοδοσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημαίνει ότι υπάρχει λογοδοσία σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, γιατί τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται άμεσα από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Και άλλωστε εμείς συναντούμε τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, στέλνουμε εκθέσεις, απαντούμε σε ερωτήματα που μας θέτουν τα εθνικά κοινοβούλια. Όλα αυτά αυξάνουν τις διαδικασίες λογοδοσίας. Και αυτό θα βελτιώσει την πρόσληψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τρόπο με τον οποίο την αντιλαμβάνεται ο Ευρωπαίος πολίτης. Είναι βασικό οι εθνικές κυβερνήσεις να έχουν την ιδιοκτησία των μεταρρυθμίσεων πράγματι και των προτάσεων που συζητώνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να τις υπερασπίζονται στα εθνικά κοινοβούλια έτσι ώστε να είναι πιο άμεση η σχέση μεταξύ αυτών που αποφασίζονται εδώ στις Βρυξέλλες, στη Φραγκφούρτη, στο Στρασβούργο και αυτού που αποκαμίζουν ως συνέστηση οι, οι πολίτες στις πατρίδες τους. Δηλαδή, όποια και αν είναι η μορφή της οριστικής συμφωνίας και καταλαβαίνω και κατανοώ τις ανησυχίες όσων ε, είναι υπέρ της συνέχισης της ε, ομοφωνίας για τη λήψη των αποφάσεων. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να έχουμε μηχανισμούς που να είναι αποτελεσματικοί, που να μπορούν να ανταποκριθούν, να δράσουν. Και η ομοφωνία λειτουργεί. Ε, οι κανόνες της ομοφωνίας συμφωνίας για ορισμένες αποφάσεις δίνουν εργαλεία που δίνουν χώρο για να χρησιμοποιηθούν με εσφαλμένο τρόπο, με ε, κακό τρόπο. Εάν ε, επικρατεί μόνο ομοφωνία, τότε ενδεχομένως πρέπει να δημιουργήσουμε θεσμικά όργανα πιο ευέλικτα για να μπορούν να λειτουργήσουν ε, ε, πιο γρήγορα. Γιατί αν τελικά συζητούμε και συνεχώς συζητούμε, όταν έρθει το πρόβλημα θα έχουμε τελικά κολλησιεργήσει. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Όταν μιλούμε για τις χρηματαγορές, η ταχύτητα είναι το στοιχείο κλειδί. Αν δεν μπορούμε να μιλήσουμε γρήγορα τότε και να δράσουμε γρήγορα, ε, τότε δεν θα έχει κανένα νόημα. Να καθορίσουμε λοιπόν τους κανόνες ξεκάθαρα, να τους συμφωνήσουμε με ομοφωνία, αλλά μετά ο μηχανισμός να λειτουργεί και να μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και όταν ε, κάποια χώρα ενδεχομένως διστάζει για δικούς της ιδιωτελείς ίσως λόγους. Και αυτό θα ήταν εξαιρετικά επιβλαβές για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σιγά σιγά προχωρούμε προς το κλείσιμο της ε, δεύτερης πρωινής συνεδρίας να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Πρώτον, είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό στο οποίο έχουμε εστιάσει και πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Γκουαλτιέρη και ο υποφαινόμενος πήραμε τη σωστή απόφαση να είναι αυτό το θέμα της συζήτησης, ο ρόλος των κοινοβουλίων κατά τη διαδικασία μετάβασης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας προς το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε όλοι πώς θα φροντίσουμε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μέλλον της Ευρώπης. Πώς να γίνει καλύτερο. Θέλουμε ασφαλέστερη οικονομία. Θέλω όμως να τονίσω τα τέσσερα βασικά εξής σημεία. Πρώτον, χρειάζεται αμοιβαία κατανόηση. Δεύτερον, χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη. Τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να εμπιστεύονται το ευρωπαϊκό το Κοινοβούλιο και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και εμείς θα πρέπει να εμπιστευόμαστε εσάς, τα Εθνικά Κοινοβούλια. Τρίτον, διαφάνεια. Να μην γίνεται τίποτε παρασκηνιακά και κλεισμένων των θυρών. Να είναι όλα διαφανή. Και τέταρτον και εξίσου σημαντικό, αποτελεσματικό της. Θέλουμε να πετύχουμε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα στην πράξη. Εάν υπάρξει αποτελεσματικότητα, μπορούμε να προσδοκούμε ότι οι μελλοντικέ μας συζητήσεις θα συνεχιστούν. Πιστεύουμε ότι στο Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να οργανωθούν συζητήσεις με τη συμμετοχή όλων. Όλους θα τους προσκαλέσουμε, όσους έχουν καλή ε, διάθεση και πίστη και μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτή τη συζήτηση για μια καλύτερη Ευρώπη. Είμαστε ακόμη στα προκαταρκτικά στάδια. Ας μην φοβούμαστε να προχωρήσουμε μαζί. Ήταν μεγάλη μου τιμή να διευθύνω αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον πρόεδρο Γκουαλτιέρη για τη συνεισφορά του, τον κύριο Μπράκμαν, την κυρία Αλμπουκέρκη και εκ μέρους της κυρίας Στογιάνοβα, της συμπροέδρου αυτής της ε, συνεδρίασης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες και όλες τις συμμετέχουσες, ιδίως όσους πήραν το λόγο. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ ε, όλους και τη γραμματεία μας και το προσωπικό της Επιτρο... των Επιτροπών μας και είναι μεγάλη μου χαρά να αναγγείλω το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Το γεύμα. Καλή σας όρεξη.